Good morning, colleagues. Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Σημείο 7 της ημερήσιας διάταξης. Ε, υποστήριξη της ε, καινοτομίας μέσω πρόληψης της ανέντιμης αποκάλυψης μυστευτικών επιχειρηματικών πληροφοριών προστασία τη τεχνογνωσία και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν αποκαλύπτονται κατά της παράνομης απόκτησης, χρήση και αποκάλυψή του. Ο κύριο Ζόμπερ Κεβίν από τη Γενική Διεύθυνση Αστερική αγορά ε, είναι εκπρόσωπο Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προ το παρόν, λέει. Ε, ε, ο, καλεσμένο μα μας είναι τμηματάρχη του τμήματο για την καταπολέμηση τη παραποίηση και τη πειρατεία. Η Επιτροπή μας αποφάσισε να συντάξει γνωμοδότηση για το, για το σχετικό νομοθέτημα με αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή στην 7η Κοινοβουλευτική Θητεία, τη Νομική Επιτροπή. Ήταν το δικαίωμα πρωτοβουλίας που άσκησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά το τέλος της θητείας της, αλλά δεν υπάρχει διαφορά, δεν υπάρχει συνέχεια και εμείς αποφασίσαμε να αφήσουμε τη γνωμοδότηση ως έχει. Μισελ Ριβαζή είναι από τους πράσινους συντάκτερες της γνωμοδότησης. Δεν έχει έρθει ακόμη όμως. Κύριος ή κυρία, κυρία, κυρία Μισελ Ριβαζή. Η κυρία Μισελ Ριβαζή διορίστηκε συντάκτηρα της γνωμοδότησης και ζητήσαμε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας κάνει μια παρουσίαση γιατί θέλουμε να είμαστε ενήμεροι για το θέμα αυτό και είναι πολύ σημαντικό για να ετοιμάσουμε το έδαφος και να μπορέσουμε να συντάξουμε μια περιστατωμένη γνωμοδότηση για το θέμα αυτό. Παρακαλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει την παρουσίασή της ε, χωρίς να ξεπεράσει το δεκάλεπτο. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Θα προσπαθήσω να περιοριστώ στο δεκάλεπτο και παρακαλώ διακόψτε με αν το ξεπεράσω. Θα το φροντίσω μην ανησυχείτε, λέει ο Πρόεδρος. Καταρχήν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή σας θα γνωμοδοτήσει για το κείμενο αυτό, γιατί πιστεύουμε ότι μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο προκειμένου να βελτιωθούν οι επιδόσεις μας σε θέματα καινοτομία ιδιαίτερα στην εσωτερική αγορά. Είναι πολύ σωστό λοιπόν και η δική σας Επιτροπή Ήτρε θα συντάξει γνωμοδότηση. Τι είναι τα εμπορικά ε, μυστικά, τα εμπορικά απόρριτα. Τεχνογνωσία ουσιαστικά. Περί αυτού πρόκειται. Κάθε επιχείρηση, άσχετα με το μέγεθός της, ε, στηρίζει την ανταγωνιστικότητά της στην τεχνογνωσία της. Και το θέμα που μας αφορά και θα σας το εξηγήσω ε, είναι ένα θέμα που αφορά ολόκληρη τη βιομηχανία και βρίσκεται στην καρδιά της οικονομίας. Τα εμπορικά απόρριτα ε, συμβάλλουν και στην καινοτομία του δικτύου και στην ε, έρευνα που είναι αντικείμενο συνεργασίας και η κοινή διαχείριση των εμπορικών απορρίτων μεταξύ εταίρων είναι το θεμέλιο της ανάπτυξης ε, συνεργειών και δικτύων καινοτομία. Όλα αυτά, επαναλαμβάνω, βρίσκονται στην καρδιά της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας μας. Το πρόβλημα που γνωρίζει ο κλάδος είναι οι απειλές. Κυρίως εξαιτίας της ανέντιμης αποκάλυψης εμπιστευτικών επιχειρηματικών πληροφοριών, γιατί δεν πρόκειται για αποκλειστικό δικαίωμα η κλοπή και η ανέντιμη αποκάλυψη ε, η χρήση εμπορικών απορρίτων είναι ένα φαινόμενο που παρουσιάζει ανωδική πορεία. Και εμείς κάναμε πολλές προπαρασκευαστικές εργασίες, το βλέπετε και στη μελέτη αντικτύπου που έχουμε επισυνάψει στην πρόταση. Και έχουμε εδώ χαρακτηριστικά παραδείγματα της βιομηχανίας από όλους τους τομείς. Μία στις πέντε εταιρείε έχει πληγεί από απόπειρα ή ουσιαστική υπεξαίρεση των εμπορικών της ε, απορρίτων την περασμένη δεκαετία και μάλιστα η τάση αυτή αυξάνεται. Και μία εταιρεία συμβούλων, η Associates, ε, μας λέει ότι μεταξύ 2012 ε, και 2013 είχαμε αύξηση από το 18% στο 25%. Το φαινόμενο αυτό αυξήθηκε και πλήττει τη βιομηχανία όλο και περισσότερο. Το πρόβλημα επηρεάζει και την εσωτερική αγορά, γιατί οι ισχύουσες εθνικές νομοθεσίες έχουν κενά. Βλέπετε εδώ τα βασικά στοιχεία που θα πρέπει να υπάρχουν για να αντιμετωπιστεί το θέμα της υπεξαίρεσης αυτών των εμπιστευτικών πληροφοριών. Βλέπετε τα κενά που δείχνει που λείπει η σχετική νομοθεσία. Δεν υπάρχει, για παράδειγμα, σαφής νομικός ορισμός στο αστικό δίκαιο για το τι εστί επιχειρηματικό ε, ή εμπορικό απόρριτο. Δεν υπάρχει καν ορισμός σε πολλά κράτη-μέλη. Οπότε υπάρχει Κανονιστικό ή νομοθετικός κατακαιρματισμό για το θέμα αυτό στην εσωτερική αγορά. Όπως είπα και προηγουμένω, οι επιπτώσει αυτή τη έλλειψη και αυτών των κενών είναι κατά τη γνώμη και κατά τη γνώμη των μελετητών μία αρνητική επίπτωση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας. Και μάλιστα τα ενάψματα για καινοτόμα διασυνοριακή δραστηριότητα μειώνονται. Και βλέπετε στα δεξιά στο κόκκινο τμήμα, 40% των ευρωπαϊκών εταιριών δηλώνουν ξεκάθαρα ότι προστιμούν να μην μοιραστούν τα εμπορικά τους απόρριτα με εταίρους από άλλα κράτη-μέλη, γιατί υπάρχει έλλειψη ασφάλειας δικαίου εξαιτία του κανονιστικού κατακαιρματισμού. Και από τις δημόσιες διαβουλεύσεις που ξεκινήσαμε διαπιστώσαμε ότι α, πάνω από το 50% των επιχειρήσεων που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο κρίνουν ότι οι διαφορές ε, στα εθνικά δίκαια καθιστούν λιγότερο ελκυστικές τις διασυνοριακές ε, δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. Οπότε από άποψη εσωτερικής αγοράς θα έπρεπε οι επιχειρηματίες να μπορούν να ζητούν οπουδήποτε μέσα στην ε, εσωτερική αγορά εταίρους. Τώρα αναγκάζονται να περιορίζονται στα εθνικά του σύνορα εξαιτία αυτής της κανονιστικής και νομοθετικής ε, αποσπασματοποίησης που υπάρχει. Τώρα, ποιος είναι ο στόχος της οδηγίας. Ο στόχος ε, ο πρωταρχικός είναι η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων και η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της νομικής προστασίας των εμπορικών απορρίτων κατά της ε, κατάχρησης ή της ε, επεξαίρεσης στην εσωτερική αγορά και να δοθούν περισσότερα ενάψματα για συνεργασίες διασυνοριακές σε θέματα ανάπτυξης, ε, έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και άρα αύξηση και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Επαναλαμβάνω, τα εμπορικά απόρριτα καλύπτουν όλους τους κλάδους, όλους τους τομείς της βιομηχανίας, ακόμη και μη τεχνολογικά προηγμένους τομείς, όπως στον τομέα των υπηρεσιών. Δίκτυα τελειών, για παράδειγμα, franchising. Και εκεί υπάρχει κοινή διαχείριση μυστικών, ε, τέτοιων εμπορικών απορρίτων, ε, επιχειρησιακά μοντέλα, επιχειρηματικά συγγνώμη μοντέλα. Και έτσι δημιουργούνται δίκτυα μεταξύ των επιχειρήσεων με κοινή διαχείριση των εμπορικών απορρίτων. Αν δεν υπάρχει ενιαία εσωτερική αγορά, δεν είναι ελκυστική μια τέτοια ανταλλαγή. Θέλουμε να μπορούν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, να ανταλλάσσουν πληροφορίες. Επαναλαμβάνω, αυτό το φαινόμενο δεν αφορά μόνο τις ε, επιχειρήσεις ε, που χρησιμοποιούν υψηλή τεχνολογία, προηγμένη τεχνολογία, αλλά όλους τους οικονομικούς κλάδους. Δεν πρόκειται να εναρμονίσουμε εδώ το ποινικό δίκαιο. Αυτό το δηλώνω κατηγορηματικά. Στο κίτρινο βέλος αναφέρεται ότι μία από τις από τους στόχους της ανακοίνωσης ε, θα ήταν να αφιπνίσουμε τα κράτη-μέλη ότι θα πρέπει να τροποποιήσουν την νομοθεσία τους. Η, πρόταση που προβάλλουμε είναι συνεκτική και με τα TRIPS, δεν ε, ενισχύει τα TRIPS. Και τα TRIPS προβλέπουν 20 ετή προστασία κατά της ανέντιμης αποκάλυψης ή κατάχρησης. Τώρα τα κράτη-μέλη προσπαθούν να μεταφέρουν αυτό το, αυτή τη διάταξη. Βέβαια και εδώ είναι κατακαιρματισμένη η εφαρμογή και δεν πιστεύουμε, και αυτό φαίνεται και στη μελέτη επιπτώσεών μας, ότι αρκούν συστάσεις προς τα κράτη-μέλη για να αλλάξει η κατάσταση. Γι' αυτό και προτείνουμε τελικά οδηγία, μία οδηγία για την εναρμόνιση του αστικού δικαίου, της προστασίας που χορηγεί το αστικό δίκτυο, ώστε να υπάρχει δυνατότητα νομικής αποκατάστασης κατά τέτοιων φαινομένων. Και στόχος είναι η βελτίωση το, της διασυνοριακής εταιρικής σχέσης. Είναι θέμα εσωτερικής αγοράς και γι' αυτό και η νομική βάση για την οδηγία αυτή είναι νομική βάση της εσωτερικής αγοράς. Θα επεκταθώ στις λεπτομέρειες ε, όταν θα απαντήσω σε ερωτήσεις. Γενικά, να δούμε το πεδίο εφαρμογής. Η οδηγία αυτή, επαναλαμβάνω, δεν αφορά την προστασία των εμπορικών απορρίτων. Γιατί μερικοί συγχαίουν ε, τα δύο θέματα. Η οδηγία αφορά την προστασία κατά της ανέντιμης αποκάλυψης εμπιστευτικών πληροφοριών ή εμπορικών απορρίτων. Καταρχήν πρέπει να δούμε τι εστί εμπορικό απόρριτο είναι ε, σχετικά ευρύ ορισμό. Καταρχήν περιλαμβάνει τι διεθνεί διατάξει των TRIPS. Ε, ορίζουμε τι εστί ανέντιμη αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών και έχετε το κόκκινο κουτί που ε, περιλαμβάνει τα στοιχεία αυτής της διάταξης και λέμε πρώτα τι δεν εστί ε, τέτοια αποκάλυψη, πιστευτικό, ανέντιμη αποκάλυψη. Η αντίστροφη ε, επινόηση ή η ανεξάρτητη ταυτόχρονη εφεύρεση δεν συνιστά ανέντιμη αποκάλυψη πληροφοριών, γιατί μπορεί δύο επιχειρήσεις να έχουν λάβει ίδιες πληροφορίες ε, και δεν έχουμε εδώ αποκλειστικά δικαιώματα. Δεν πρόκειται για πνευματική... Είναι ένα είδος πνευματικής ιδιοκτησίας, αλλά όχι αποκλειστικό δικαίωμα. Ένα άλλο στοιχείο του άρθρου 2 είναι οι εξαιρέσει πότε και υπό ποιου όρου ένα εμπορικό απόρριτο, για λόγους δημοσίου συμφέροντος για παράδειγμα, να αποκλειστεί. Αυτό αναφέρεται στο σημείο 2, στην παράγραφο 2. Ορίζουμε λοιπόν το πεδίο εφαρμογής στην οδηγία και μετά προβλέπονται τα ένδικα μέσα. Οι προσφυγές σε περίπτωση που λάβει η χώρα μια τέτοια κατάχρηση, ανένδυμη αποκάλυψη, υπεξαίρεση. Έχουμε κάποια ασφαλιστικά μέτρα, ε, μέτρα για τα συγκεκριμένα προϊόντα που εμπίπτουν σε αυτό το εμπορικό πόρυτο. τα προϊόντα της παραβίασης και εδώ προβλέπεται και προσωρινή κατάσχεση και προβλέπουμε και κάποια αναλλακτικά μέσα, αναλλακτικά σε σχέση με τα ασφαλιστικά μέτρα. Ένα τρίτο μέρος μπορεί καλή την πίστη να έχει στην κατοχή το ένα εμπορικό απόρριτο που ίσως τύχει κατάχρηση. Αυτό μπορεί να το αφισβητήσει μια επιχείρηση. Αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Και ο δικαστής θα πρέπει να έχει δικαίωμα να επιδικάσει εναλλακτικά μέτρα αντί να επιβάλλει ασφαλιστικό μέτρο για την απαγόρευση της χρήσης του προϊόντος ή την απαγόρευση της χρήσης του εμπορικού απορρίτου. Αποζημιώσεις και δημοσίευση των αποφάσεων επίσης προβλέπονται στην οδηγία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις ασφαλιστικές δικλίδες, δύο είναι τα σημαντικά εδώ. Το ένα, το γεγονός ότι καμία εταιρεία δεν μπορεί σε ανοιχτό δικαστήριο να υποβάλει προσφυγή. Για προφανείς λόγους. Γιατί σε μια ανοιχτή δίκη αποκαλύπτεται εμπορικό απόρριτο. Μάλιστα, όλος παραδόξως σε μερικά κράτη-μέλη δεν υπάρχει τέτοια εγγύηση να υπάρχει ένα τέτοιο όριο για να μην δημοσιεύονται ουσιαστικά αυτά τα εμπορικά απόρριτα, να γίνεται δηλαδή ανταλλαγή πληροφοριών πολύ περιορισμένα μεταξύ των, επι... Ε, των αντιδίκων μόνο και όχι σε μία ανοιχτή δίκη. Ή υπάρχει νομοθετική διάταξη και δεν χρησιμοποιείται ακόμα σε κάποια κρατημέλη. Διασφάλιση της εμπιστευτικότητας ε, είναι σημαντικό στοιχείο του κειμένου που προβλέπεται στο άρθρο 8. Αν θέλετε μπορούμε να επισέλθουμε σε λεπτομέρειες. Κάτι άλλο. Και επανέρχομαι σε αυτό γιατί δεν είναι αποκλειστικό δικαίωμα, το τονίζω αυτό. Και φροντίσαμε γιατί πιστεύουμε αν και το Κοινοβούλιο θα απαντήσει, ότι βρήκαμε τη σωστή ισορροπία. Δηλαδή αφενός ε, θεσπίσαμε κάποιες ασφαλιστικές δικλίδες με βάση την αρχή της αναλογικότητας, ώστε να μην είναι δυσανάλογα τα μέτρα σε σχέση με την κατάχρηση, αλλά και να περιορίσουμε τον κίνδυνο της κατάχρησης ή της υπεξαίρεσης. Γιατί μία επιχείρηση δεν μπορεί μετά από δύο χρόνια να ισχυριστεί ότι α, κάποια εταιρεία καταχράστηκε το εμπορικό μου απόρριτο θα προσφύγω, γιατί συχνά κάποιοι εργαζόμενοι εγκαταλείπουν μια εταιρεία, έχουν μια ιδέα για το έργο της εταιρεία, το οποίο δεν συνεχίστηκε από την εταιρεία, μετά ανοίγουν τη δική τους επιχείρηση και αναπτύσσουν περαιτέρω μια ιδέα. Βέβαια, πολύ συχνά η νέα επιχείρηση είναι ο καλύτερος πελάτης της πρώτης επιχείρησης. Αν πάνε όλα καλά. Αλλά μπορεί η πρώτη εταιρεία μετά τρία-τέσσερα χρόνια να προσπαθήσει να αναχαιτήσει την εξέλιξη της δεύτερης εταιρεία και να επικαλεστεί κατάχρηση των αρχικών πληροφοριών που αποτέλεσαν τη βάση για την ανάπτυξη της καινοτομίας από τη δεύτερη εταιρεία. Γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχει περιορισμός. Και από τη στιγμή που κάποιο ε, θεωρεί ότι έγινε υπεξαίρεση ενό εμπορικού απορρίτου θα πρέπει να ισχύει μια προθεσμία διετής για το δικαίωμα προσφυγής. Τώρα, έχουμε και κάποια δικονομικά μέτρα. Ποια είναι τα ωφέλη της οδηγίας. επαναλαμβάνω, καλύτερη διασυνοριακή προστασία των επιχειρήσεων που θα οδηγήσει σε ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και σε πιο αποτελεσματικά δίκτυα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, περισσότερη συνεργασία και καινοτομία. Και άρα αύξηση ε, της ανταλλαγής ε, ε, εμπορικών πληροφοριών και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ε, επιχειρήσεων που συνεργάζονται μεταξύ τους και βελτίωση της καινοτομίας και της εσωτερικής αγοράς γενικώ. Τώρα, ποια ήταν τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης που οργανώσαμε. Βλέπετε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και αυτό είναι ενδιαφέρον, θα σας πω ειλικρινά τι πιστεύω και μετά θα απαντήσω σε ερωτήσεις. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που σας διαβεβαιώ γιατί και εγώ για 20 χρόνια παρακολουθώ τα θέματα εσωτερικής αγοράς, είναι απρόθυμες. Ε, φοβούνται οποιαδήποτε μορφή νέας νομοθεσία γιατί φοβούνται το γραφειοκρατικό άχθος. Στην περίπτωση αυτή όμως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι αναφαντών υπέρ ευρωπαϊκής νομοθεσίας για το θέμα αυτό. Επίσης, οι πολίτες φαίνεται ότι δεν ενδιαφέρονται. Δεν θεωρούν ότι είναι απαραίτητη μια τέτοια ρύθμιση. Πολλοί πολίτες που έλαβαν μέρος στη διαβούλευση φάνηκε ότι δεν κατάλαβαν περί την όσο Δεν λέω ότι όλοι θα έπρεπε να συμφωνούν, αλλά φαίνεται ότι δεν κατάλαβαν περί την πρόκειται. και θα πρέπει να γίνει και εδώ στο Κοινοβούλιο ευρυθή συζήτηση. Εμείς βρήκαμε, θεωρούμε ότι βρήκαμε τη σωστή ισορροπία, αλλά εσείς θα το κρίνετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα θα έχουμε ε, τον γύρο των, ε, αντιπροσω... των εκπροσώπων των ε, πολιτικών ομάδων. Ο κύριος Ρίβαση από τους Πράσινους. Η κυρία Ρίβαση από τους Πράσινους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ για αυτή την παρουσίαση. Όντως, όπως είπατε κι εσείς, η οδηγία αυτή απορρά ε, την απόκτηση, ε, δημοσιοποίηση εμπορικών μυστικών και θέλουν και ε, κάποια μέτρα προκειμένου να διορθωθεί η κατάσταση. Ο ορισμός καταρχάς ε, του εμπορικού μυστικού είναι βασικός εδώ. Περιλαμβάνει τρία στοιχεία. Οι πληροφορίες πρέπει να είναι εμπιστευτικές, περιλαμβάνουν κάποια στοιχεία λόγω ακριβώς του απορρίτου και ε, το εμπορικό ε, απόρριτο έχει τύχει κάποιων συγκεκριμένων μέτρων από τον κάτοχο του μυστικού αυτού. Θεωρώ ότι ο ορισμός αυτός είναι πάρα πολύ ευρύς και δίνει περιθώριο για πολλές ερμηνείες και πολλές ασάφειες. Ε, ενώ κανονικά εμείς θέλουμε να έχουμε ακριβώς το αντίθετο. Εγώ θα προτιμούσα λοιπόν έναν ε, ε, ορισμό των εξαιρέσεων, πια δεν προβλέπονται από αυτή την οδηγία, ε, παραδείγματος χάρη εμπορικά απόρριτα για την δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Ε, αυτό το οποίο θα μπορούσε να συμβεί είναι ότι όλα τα οποία πιθανόν μπορεί να έχουν ένα εμπορικό χαρακτήρα θα πρέπει να είναι απόρριτα, να προστατεύονται και επομένως θα πρέπει να έχουμε προστασία δυσανάλογη. Ε, και εδώ όλα προκύπτουν από τον ορισμό αυτού που αποκαλείται εσείς εμπορικό απόρριτο. Καταρχάς η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται πολύ καλά από τα συστήματα των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και επομένως θέλουμε να έχουμε και ένα ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Αν υπάρχει κάποιο απόρριτο ε, μιας ε, μεταπτυχιακής βιομηχανίας υπάρχει δυνατότητα διπλώματος ευρεσιτεχνίας και υπάρχουν και άλλα εργαλεία και αυτό είναι η τεχνογνωσία. Παραδείγματο χάρη, στι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν εμπορικό απόρριτο, αλλά εμεί προστατευόμαστε πάρα πολύ καλά από την νομοθεσία μα. Έχουμε τα διπλώματα ευρεσιτεχνία και έχουμε και την τεχνογνωσία. Και οι επιχειρήσει μπορούν κάλλιστα να εφαρμόζουν την νομοθεσία. Και αν δεν υπάρχει κάτι σε μια χώρα, τότε θα πιέσουμε ώστε να εφαρμοστούν και αυτά. Να υπενθυμίσουμε επίση ότι το δίπλωμα ευρεσιτεχνία είναι ένα στοιχείο κλειδί το οποίο βοηθά τι επιχειρήσει να προχωρήσουν την καινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη. Το δίπλωμα ευρεσιτεχνία επιτρέπει στον κάτοχο να ε, μην επιτρέψει οποιαδήποτε χρήση, πώληση και ούτω καθεξής χωρί την σύμφωνη γνώμη τη. Και οι επιχειρήσεις ε, πρέπει να κάνουν επενδύσει απαραίτητε για την καινοτομία. Αντίθετα με το εμπορικό απόρριτο, όπω παρουσιάζεται εδώ στο κείμενο, το δίπλωμα ευρεσιτεχνία επιτρέπει να προστατεύουν πούμε, προστατεύοντας ταυτόχρονα και την καινοτομία. Και ε, δεν επιτρέπεται η δημοσίευση των στοιχείων όσον αφορά την καινοτομία. Πώς μπορούν λοιπόν να ε, δεχτούμε ότι δεν θα μπορούμε να έχουμε καλύτερες βελτιώσεις αν δεν υπάρχει καμία νομική πρόσβαση σε δυνατότητες καινοτομίας. Τα εμπορικά απόρριτα δεν θα πρέπει να είναι μια έννοια η οποία στόχο έχει ε, να μπορέσει να ε, χρησιμοποιήσει της αποτυχίας των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας είναι ουσιαστικά ένα κοινωνικό συμβόλαιο που επιτρέπουν να ε, προχωρήσει η καινοτομία. Το να προσθέσουμε το εμπορικό απόρριτο εδώ δεν αποτελεί λύση ούτε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ούτε για την κοινωνία. Ε, Και αν δω τα στοιχεία της έρευνά σας, αυτό το οποίο βλέπω περισσότερο είναι ότι αυτοί οι οποίοι είναι περισσότερο αντίθετοι είναι οι πολίτες στο εμπορικό απόρριτο. Υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία προστατεύονται από την νομεσία, νομοθεσία, όπως για παράδειγμα το άρθρο 30 της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων για τις ε, ε, αδικαιολόγητες ε, απολύσεις και το δικαίωμα στην υγεία. Ε, για λόγους υγείας, για παράδειγμα, το εμπορικό απόρριτο θα πρέπει να προστατεύεται γιατί θα πρέπει οι επιχειρήσεις να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους και πρέπει να προστατεύεται η καινοτομία και οι πολίτες. Και έχω ένα παράδειγμα να σας δώσω εδώ. Δείτε για παράδειγμα τι γίνεται με το σχιστολιστικό φυσικό αέριο. Έγινε ολόκληρη διαμάχη εναντίον των αμερικανικών επιχειρήσεων, διότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις δεν θέλουν να μας δώσουν τον τύπο ε, αυτού του κοκτέιλ των χημικών, προϊόν για την, ε, χημικών προϊόντων για το σχιστολιθικό φυσικό αέριο. Μπορεί αυτό να θεωρηθεί εμπορικό απόρριτο. Εμείς όμως έχουμε νομοθεσία βάσει του ΡΙΤΣ η οποία υποχρεώνει τον ε, παραγωγό να δώσει τη χημική σύνθεση γιατί μπορεί να περιλαμβάνει τοξικές ουσίες που δεν επιτρέπονται. Εγώ λοιπόν σας ε, ε, ομολογώ ότι αυτό το εμπορικό απόρριτο μου δημιουργεί προβλήματα διότι δεν είναι ακριβώς ε, ακριβής ο ορισμός, δεν ξέρουμε τι θα περιλαμβάνεται και υπάρχουν κάποιες επιχειρήσεις που θέλουν να το εκμεταλλευτούν αυτό ώστε να μην δίνουν πληροφορίες στην κοινωνία. Επιπλέον, αναγνωρίζω ότι η κοινωνία της γνώσης ε, ε, δεν θέλει να έχει κατάχρηση εμπιστευτικών πληροφοριών και θέλει να βοηθήσει τις επιχειρήσεις στην ανταγωνιστικότητα και ελπίζω ότι υπ' αυτό το πνεύμα προτάθηκε συγκεκριμένη οδηγία. Έχω κάποιες αμφιβολίες βέβαια που θα σας εξηγήσω αργότερα. Ε, σας παρακαλώ ολοκληρώστε διότι μιλάτε πάνω από πέντε λεπτά κυρία Ριβαζή. Ζητώ συγγνώμη. Termine. Apparemment, και ολοκληρώνω. Οι Διατλαντικέ συμφωνίες και αυτές ε, πλήττονται από το θέμα του εμπορικού απορρίτου γιατί το είδα αυτό στις διατλαντικές συμφωνίες. Διότι δεν επιτρέπεται η δημοσιοποίηση σημαντικών πληροφοριών. Ε, θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μου αποδείξει για ποιο λόγο ε, χρειαζόμαστε ένα τέτοιο κείμενο για να προστατεύσουμε την καινοτομία στην Ευρώπη. Διότι αν δω τη μελέτη επιπτώσεων δεν βρήκα πουθενά κάτι τέτοιο και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χρειάζομαι επιχειρήματα που να μου πούνε ότι αν ε, προχωρήσει αυτή η νομοθεσία θα μπορέσουμε να προωθήσουμε την καινοτομία. Για του κοιόδη συζητητέ προτείνω τρία λεπτά γιατί πρέπει να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα. Ο κύριο Πατριτσέλο του ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στον τομέα της επιστήμης και της καινοτομίας η Ευρώπη βρίσκεται στην πρώτη γραμμή και έχει τις δυνατότητες ε, να γίνει παγκόσμιος ηγέτης. Γι' αυτό ακριβώ και θα πρέπει να βελτιώσουμε τι προποθέσει βάσει των οποίων οι επιχειρήσει διεξάγουν τι καινοτόμε δραστηριότητέ του και πιο συγκεκριμένα μέσω προστασία των επενδύσεων όσων επενδύουν στη γνώση μειώνοντας το κόστος ε, του κατακαιρματισμού της αγοράς, ε, της ενιαίας αγοράς και κάνοντας μια Ευρώπη ένα ε, όρο που θα ε, πρημοδοτεί την καινοτομία. Θεωρούμε ότι αυτά είναι ένα απόσπαστο στοιχείο της πολιτικής καινοτομίας, διότι επιτρέπουν στους ανθρώπους που καινοτομούν να έχουν μέσα, ε, ο, μέσω των οποίων να βλέπουν τα αποτελέσματα ε, των όσων έκαναν και ταυτόχρονα προσφέρουν και τα απαραίτητα κίνητρα για να επενδύσουμε σε νέες επενδύσεις ε, ε, για το μέλλον. Παρά το γεγονός ότι δεν είναι κλασικά πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά, ο απόρριτο ή κάποιοι τύποι παρασκευής, νέες ουσίες και υλικά, τεχνολογίες που ακόμα δεν την χάνουν διπλώματος ευρεσιτεχνίας και επιχειρηματικά απόρριτα, είναι αναπόσπαστο στοιχείο για να μπορέσουμε να ε, προστατεύσουμε την ε, πνευματική κληρονομιά που είναι βασικός μοχλός της επιχειρηματικότητας και της γνώσης. Τα εμπορικά απόρριτα λοιπόν θεωρούνται στρατηγική σημασία για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία. Αν δεν υπάρχει κατάλληλη προστασία ή είναι λυπής η προστασία, τότε θα έχουμε αρνητικές συνέπειες για τις ε, στρατηγικές καινοτομίας των επιχειρήσεων. Η παγκοσμιοποίηση η ε, εξωτερήκευση των αλυσίδων ε, διανομής σημαίνει ότι το εμπορικό απόρριτο μπορεί ε, να κλαπεί ανα πάσα στιγμή και μπορεί φυσικά οι μέθοδοι παραγωγής να αντιμετωπίζουν προβλήματα, γι' αυτό και χρειαζόμαστε μεγαλύτερη προστασία, ενισχυμένη προστασία εντός της εσωτερικής αγοράς, όπου αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κατακαιρματισμένο πλαίσιο με μεθόδους οι οποίες ε, πολύ συχνά αποθαρρύνουν, ιδίως όταν υπάρχουν ε, διαφιλονικίες και επίμαχα σημεία μεταξύ των επιχειρήσεων. Το να υπάρχει ένα εναρμονισμένο πλαίσιο με κανόνες οι οποίοι θα είναι σαφείς σημαίνει ότι διασφαλίζουμε την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και βελτιώνουμε την αποδοτικότητά τους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ συνάδελφε και εξ ονόματος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών ως και η η κυρία Βέρνερ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώ ορίζω την πρωτοβουλία επί της αρχής και ιδιαιτέρω για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για δεδομένα βάση επιστημονικών δεδομένων έχει μεγάλη σημασία. Αλλά δυστυχώς οι επιχειρήσεις αυτές δεν έχουν τις δυνατότητες να προστατεύσουν επαρκώς τα δεδομένα αυτά. Και η πιο έντονη ψηφιοποίηση, η κατανομή και η ανάθεση τέτοιων συμβατικών υποχρεώσεων αυξάνουν τις ε, απαιτήσει. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να είναι πιο έντονη η συνεργασία διασυνοριακή σε θέματα τέτοιων στοιχείων. Γι' αυτό λοιπόν καλό είναι σε πανευρωπαϊκό επίπεδο να υπάρχει και μια ασφάλεια δικαίου. Να κάνω και κάποιες άλλες παρατηρήσεις για κάποια σημεία τα οποία θεωρώ ότι θα πρέπει να τα συζητήσουμε ακόμη. Γιατί κατά πρώτον αυτή η οδηγία δεν μπορεί να είναι λευκή επιταγή σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια και να αποβεί εις βάρος των καταναλωτών και σε ό,τι αφορά ενδεχόμενες καταχρήσεις. Θα πρέπει να προφυλαχθούμε. Κατά δεύτερον, σε ό,τι αφορά τον ορισμό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει να κάτσουμε να σκεφτούμε κατά πόσον οι πληροφορίες οι οποίες ενδεχομένως να είναι εμπορική αξίας θα πρέπει να συμπεριληφθούν ή όχι. Και τρίτον, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι και οι εργαζόμενοι σε ό,τι αφορά καταχρήσεις θα μπορούν να αναφερθούν, να στραφούν προς ένα συνδικάτο χωρίς να έρθουν σε αντίθεση με τις διτάξεις της οδηγίας. Οποιαδήποτε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα υπόκειται στην οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και οι ΕΠΑ φαίνεται ότι ζητούν μια τέτοια ρύθμιση να συμπεριληφθεί στη Συμφωνία Ελευθερίου Μπορείου TTIP. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε πώς έχει η κατάσταση σήμερα και κατά πόσον υπάρχουν τέτοιες ε, συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά είναι τα σημεία που θα πρέπει να μας απασχολήσουν και προσβλέπω στη συνεργασία με την συνάδελφο Ριβάζη. Thank Σας ευχαριστώ για την ε, ομιλία σας. Ο συνάδελφος Πέτερσον, αντιπρόεδρος. Αντικαθιστά τον ε, σκιώδη Φιλίπ Τεμπάκερ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίαση αυτή. Συμφωνούμε προφανώς με τον απότερο στόχο της πρότασης, που είναι η εναρμόνιση της νομοθεσίας σε κάποιο βαθμό και κατά πάσα πιθανότητα η οδηγία είναι ο πλέον ενδεδειγμένο τρόπος για να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου σε όλη την Ευρώπη. Συμφωνούμε λοιπόν επί της αρχής ότι χρειαζόμαστε καινοτομία προκειμένου να υπάρξει ανάπτυξη και θέσεις εργασίας, προκειμένου λοιπόν να επενδύσουν στην καινοτομία. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η καινοτομίε του προστατεύονται, το οποίο ελπίζουμε ότι θα οδηγήσει με τη σειρά του σε νέα προϊόντα και σε νέε επενδύσει. Σύμφωνα με τη μελέτη που προκύπτει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν δεν έχουν πάντα επαρκή μέτρα για να προστατεύσουν αυτή την καινοτομία IPR. Άρα θέλουμε να δημιουργήσουμε ασφάλεια δικαίου και να δώσουμε και ένα ελάχιστο επίπεδο συλλογικής προσφυγής στις επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Δύο ερωτήσει έχω να κάνω προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο άρθρο 7, πείτε μας ποια είναι η επιχειρηματολογία σε ό,τι αφορά την ε, περίοδο περιορισμού, σε ό,τι αφορά νομική αγωγή για ένα ε, και δύο έτη μετά από αποκάλυψη παράνομης χρήσης ε, δεδομένων. Γιατί λοιπόν γίνεται αυτό, γιατί προβλέπεται αυτό, ρωτώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και το δεύτερον, αν όντω ένα εθνικό δικαστήριο αποφανθεί ότι χρησιμοποιήθηκαν ε, εμπορικά πόρτα με παράνομο τρόπο, τι γίνεται σε ό,τι αφορά το μέλος που έχει πληγεί, σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα τα πνευματικά δικαιώματα. Ποιο θα καθορίσει τα πνευματικά δικαιώματα αυτά. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, λέει και ο Πρόεδρο. Έχουμε άλλο ένα σχόλιο από την κυρία Σάντερ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ πιστεύω ότι στην εποχή της γνώσης ε, η προστασία των δεδομένων αποτελεί θέμα στρατηγικής σημασίας για τις επιχειρήσεις. Οι μεγάλες επιχειρήσεις ε, είναι πολύ καλύτερα εξοπλισμένες και μπορούν να προστατευτούν από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πολύ αμφιβάλλουν ε, σήμερα για το τι δυνατότητες έχουν να προστατεύσουν τα δεδομένα τους. Μιλήσαμε για το δίπλωμα ευρεσιτεχνία, αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι το δίπλωμα ευρεσιτεχνία είναι το κατάλληλο σύστημα για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει, γιατί πρόκειται για μια δαπανηρή και περίπλοκη διαδικασία. Πρέπει να γίνουν μεταφράσει και ούτω καθεξή. Εγώ θα προτιμούσα μια σταθερή, στιβαρή, βέβαιη, ασφαλή ε, εύληπτη και προσιτή νομική βάση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και χρήσιμο θα ήταν ε, να εξετάσουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, να καινοτομήσουν όχι μόνο τα προϊόντα τους, αλλά να καινοτομήσουν θεσπίζοντας ε, ένα ίδιο σύστημα προστασίας δεδομένων. Ευχαριστώ. Uh, uh, Ευχαριστώ πολύ. Άλλος. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κατάλληλη προστασία των εμπορικών απορρίτων είναι θεμελιώδης σημασίας κατά την άποψή μας, κυρίως για τις μικρότερες επιχειρήσεις. Πρέπει να υπάρχει μια σαφής πολιτική για την πνευματική διοκτησία και για τα διπλώματα ευρεσιτεχνία. Και αυτό το οποίο μα εκπλήσει περισσότερο είναι το γεγονό ότι συζητούμε νομοθεσία για το θέμα αυτό, ενώ ταυτόχρονα γίνεται διαπραγμάτευση για μια συμφωνία ε, όπω η TTIP. Πώς μπορούμε να έχουμε συνέπεια μεταξύ των δύο προσεγγίσεων. Πώς μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα χάσουμε τη δέουσα ισορροπία μεταξύ αυτού το οποίο θα πρέπει να την χάνει εμπορία, επομένω να προστατεύεται από τον αθέμητο ανταγωνισμό, σε σχέση με το δικαίωμα ενημέρωσης για την προστασία των καταναλωτών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την παρατηρήσή σας. ο εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης ε, ΜΑΡΚΤ ε, να ε, πάρει το λόγο για να μας απαντήσει σε ερωτήσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ξέρω ότι καθυστέρησα πολύ, θα είμαι σύντομος, αλλά να σας πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορώ να μιλήσω με τα μέλη, την εισηγήτρια και τους βοηθείς τους. Καταρχάς, δύο λόγια όσον αφορά τον ορισμό. Κύριε Ριβαζή, θα σας μιλήσω γαλλικά. Πιστεύω ότι στην αρχή της παρουσίασης μου σας είπα ότι πρέπει να δούμε τον ορισμό. Όπως είπατε κι εσείς, όχι το τι ακριβώς είναι εμπορικό απόρριτο, αλλά το τι δεν είναι εμπορικό απόρριτο. Και αυτό περιλαμβάνεται στο κείμενο και επιπλέον α, αυτό που πρέπει να ορίσουμε είναι αυτό ε, που, είναι η παράνομη ε, χρήση, η υπεξαίρεση ουσιαστικά. Και το κείμενο είναι πολύ σαφές. Ε, αναφερθήκατε σε κάποιες περιπτώσεις στις οποίες θα υπάρχουν η νομική υποχρέωση να δίνονται τα στοιχεία και το κείμενο είναι απόλυτα σαφές. Αυτές οι νομικές υποχρεώσεις ε, υπάρχουν και δεν μπορεί κάποιος να ε, επικαλεστεί εμπορικό απόρριτο για να μην δημοσιοποιήσει αυτές τις πληροφορίες. Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ σημαντικά αυτά για τη δημόσια υγεία και για το περιβάλλον και είμαι διατεθειμένη φυσικά να το συζητήσω και μαζί σας. Ε, είναι μία κλειδί ο ορισμός και επομένως Νομίζω ότι το περιλαμβάνει αυτό ο ορισμός, αλλά είμαστε διατεθειμένοι να το συζητήσουμε μαζί σας και να τα αλλάξουμε. Επειδή δεν έχω πολύ χρόνο τώρα, να σας πω για να απαντήσω την ερώτηση για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Να σας απαντήσω γι' αυτό, γιατί νομίζω ότι η κυρία Σαντέρα αναφέρθηκε σε αυτό, θεωρώ ότι το εμπορικό απόρριτο συμπληρώνει το δίπλωμα ευρεσιτεχνία. Αυτό διαπιστώσαμε. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Μπορείτε να έχετε τα διπλώματα ευρεσιτεχνία για ένα κινητήρα ε, αεροπλάνου, αλλά ε, θα πρέπει να υπάρχει και η τεχνογνωσία για να το κατασκευάσουμε. Ε, γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να γίνεται ανταλλαγή πληροφορών μεταξύ των διαφόρων παραγόντων ώστε να μπορέσει να κινηθεί για παράδειγμα ένα αεροπλάνο. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Ένα άλλο στοιχείο είναι όπως είπατε και εσείς, πολλές επιχειρήσεις και κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν καινοτομίε οι οποίες θα μπορούσαν να προστατεύονται από ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας αλλά έχουν επενδύσει για αυτές τις καινοτομίε. Και αυτό καλύπτεται από το εμπορικό απόρριτο. Και να σας υπενθυμίσω ότι δεν πρόκειται για αποκλειστικό δικαίωμα. Ο καθής μπορεί να πάρει ένα προϊόν, να το, ε, να το εξετάσει, να δει πώς δουλεύει μηχανικά και να βρει ποιο είναι το εμπορικό απόρριτο. Ε, επομένως αυτό προστατεύει και νομίζω ότι είναι σημαντικό. Τώρα, η ερώτηση του κυρίου Πέτερσον, γιατί δύο χρόνια. Εμείς θεωρούμε ότι δύο χρόνια αρκούν δύο χρόνια από τη στιγμή που η επιχείρηση διαπιστώνει ότι υπήρξε υπεξαίρεση. Α, κατά την άποψή μας δίνει τη δυνατότητα για ένδικα μέσα εντός δύο ετών και γιατί αυτό, διότι ελοχεύει ο κίνδυνος αν υπερβούμε τη διετία η επιχείρηση ουσιαστικά μπορεί να αναλάβει δράση για να σταματήσει μια καινοτομία. Πιστεύω ότι είναι σημείο κλειδί, έχετε δίκιο, το Συμβούλιο έχει διαφορετική άποψη. Εμείς όμως είμαστε υπέρμαχοι αυτού του στοιχείου και είμαστε διεθυμένοι να το συζητήσουμε μαζί σας. Αυτή ήταν μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση και νομίζω κύριε Πρόεδρε ότι... Α, και κάτι ακόμα πώς ε, θα γίνονται, δίνονται αποζημιώσεις. Ε, προβλέπουμε αποζημίωση ε, μέσω πνευματικών δικαιωμάτων. Ε, ο δικαστής πολύ εύκολα θα μπορεί να το επιδικάσει αυτό ε, και αναπερίπτωση και όταν Αναφέρθηκε ε, και η κυρία Σάντερ στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πώς μπορούμε να τις προστατεύσουμε. Να σας πω ότι στην οδηγία αυτή έχουμε μια πολύ ε, ανεπτυγμένη διαδικασία αξιολόγησης ε, και ελέγχου. Πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις μας λένε ότι θα πρέπει να δίνονται καλύτερες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, θα πρέπει να εφαρμόζουν τα πράγματα αυτά. Όλα αυτά θα συνοδεύουν αυτή την οδηγία. Ελπίζω να πάτε σε ερωτήσεις. Όλες τις ερωτήσεις. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ζητήσω από την κυρία Ριβαζή να συνοψίσει για τη συζήτηση αυτή. Κυρία Ριβαζή, αν μπορείτε να συνοψίσετε, αν έχετε κάτι να προσθέσετε και να απαντήσετε, να διασκεδάσετε τυχόν αμφιβολίες. Έχετε το λόγο. Uh, Αν κάνω μια ανάλυση, μια ανακεφαλαίωση της συζήτησης, θα έλεγα ότι χρειαζόμαστε έναν ε, ε, ορισμό που θα είναι εύληπτος, θα μπορούν όλοι να τον ε, κατανοούν αν στόχος είναι η εναρμόνιση των διαφόρων νομοθεσιών. Επίσης είπαμε ότι θέλουμε να ευνοήσουμε την καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ακόμη και αν δεν κατέχουν δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για το τεχνικό σκέλος. Ίσως αυτό ε, συμβάλλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Αυτό ακούσαμε. Επίσης ε, θα ακολουθήσει συζήτηση για το κατά πόσο η οδηγία θα γίνει για να ενισχυθεί η καινοτομία και η ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ή μήπως θα τη χρησιμοποιήσουν για άλλους σκοπούς αυτή την οδηγία οι μεγάλες επιχειρήσεις. Νομίζω ότι μου θα ήταν και αυτή η συζήτηση να γίνει. Και φαντάζομαι ότι με τους και ηγητές ε, θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε αυτή την οδηγία. Εγώ πάντως διαβάζοντας το σχέδιο οδηγίες δεν πολύ κατάλαβα. Γιατί έχουμε ήδη κάποια μέσα νομοθετικά. Δεν βλέπω την υπεραξία αυτή τη, την προστιθέμενη αξία αυτή τη οδηγία. Θα πρέπει λοιπόν ε, να εξηγήσουμε πώς αυτή η πρόταση για το εμπορικό απόρριτο θα βελτιώσει τη λειτουργία των ε, μικρομεσαίων και άλλων επιχειρήσεων. Απευθύνω λοιπόν έκκληση προς και οδησηγητές για συνεργασία προκειμένου να βελτιώσουμε την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστούμε κύριε Ριβαζή. και ευχαριστώ και τον κύριο Ζαν Μπέζεβα από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς που μας έκανε την παρουσίαση από την Επιτροπή. Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι, προτάσεις που περιλαμβάνει η οδηγία σας προκειμένου να προστατευτούν ε, οι επιχειρήσεις ε, έναντι ανέντιμης παράνομης απόκτησης, χρήσης και δημοσιοποίησης εμπορικών ε, απορρίτων. Είναι πολύ σημαντική αυτή η προστασία της τεχνογνωσίας. Ευχαριστούμε λοιπόν και για την παρουσίαση και για τις απαντήσεις που δώσετε και θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας στο μέλλον. The next topic. Επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι ψηφοφορία, ηλεκτρονική ψηφοφορία. έχει προβληθεί για τις 10. Θα περιμένουμε λοιπόν ακόμη 4-5 λεπτά. Στις 10 ακριβώς θα αρχίσει η ψηφοφορία. Γιατί το θέμα είναι πολύ σημαντικό. Θα ψηφίσουμε για το Γενικό Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Οικονομικό Έτος 2015. Όλα τα τμήματα. Έχουμε ακόμα τρία λεπτά, γι' αυτό λοιπόν να σας ενημερώσω σε ό,τι αφορά τα... το σημείωμα που λάβαμε σε ό,τι αφορά τη χθεσινή συνεδρία των συντονιστών. Οι συντονιστές λοιπόν τι αποφάσισαν, αποφάσισαν τα εξή. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά τις ε, εκθέσεις με απλοποιημένη διαδικασία σε ό,τι αφορά τη συμφωνία για τη συμφωνία GNSS με το Μαρόκο, συμφωνία για τη συνεργασία σε θέματα επιστήμης με την Ουκρανία. Ο εισηγητής είναι πρόεδρος της Επιτροπής μας. Συμφωνήσαμε επί εκθέσεων ίδιας πρωτοβουλίας σε ό,τι αφορά τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη, ΕΛΚ. Ε, ανάπτυξη μιας βιώσιμης ευρωπαϊκής μηχανίας για βασικά μέταλλα, σοσιαλιστές και δημοκράτες, πράσινο σχέδιο δράση για τις μικρομεσαίες ε, Άλτε, φιλελεύθερη και καινοτομία σε ό,τι αφορά την μπλε οικονομία, η ΓΚΟΕ. Γνωμοδοτήσεις, η οδηγία για τα απόβλητα, Άλτε, φιλελεύθερη, Ευρωπαϊκή Δασική Στρατηγική, ECR. Αποφάσεις τώρα. Η Συντονιστέ λάμβανε και τι εξή αποφάσει. Καταρχά σε ό,τι αφορά τι αποστολέ τη Επιτροπή Ήτρα και τι ακροάσει το 2015. Θα σας τα παράσχουμε όλα αυτά ως πληροφορίες. Κατά δεύτερον, όρισαν τον Αντιπρόεδρο της Ήτρα, τον κύριο Πέτερσε, ως ε, μόνιμο ε, εισηγητή για τέτοια θέματα της Ήτρε που έχουν να κάνουν με την ισότητα των φύλων. Και τρίτον, αποφάσισαν σε ό,τι αφορά τα μέλη της Ήτρε για την ε, διαθεσμική ομάδα για το Γαλιλαίο. Και κατά τέταρτον αποφάσισαν να προετοιμάσουν και να δουλέψουν σε ό,τι αφορά το COP20 όπως και τα τελευταία χρόνια σε συνεργασία με την Επιτροπή ΕΝΒΗ. Συνεργασία λοιπόν αποφασίστηκε με την Επιτροπή ΕΝΒΗ σε ό,τι αφορά θέματα για τη διάσκεψη αλλαγή του κλίματος COP20. Τώρα, αυτές τις πληροφορίες μπορείτε να τις βρείτε και στο φάκελό σας και στο διαδίκτυο. Διατίθενται τα σχετικά στοιχεία για τις ακροάσεις των επιτρόπων τώρα. Το πιο σημαντικό θέμα που έχουμε μπροστά μας μεταξύ 29 Σεπτεμβρίου και 7 Οκτωβρίου του 2014, θα ήθελα να τονίσω ότι ως Επιτροπή βιομηχανία εξ αρχής έχουμε αναμειχθεί στη διαδικασία αυτή μέχρι και το τέλος της διαδικασίας κάθε μέρα γιατί συνολικά έχουμε 6 ημέρες 29η, 30η, η πρώτη, η Δευτέρα, Τρίτη η 6η και η 7η Οκτωβρίου. Έξι ημέρες λοιπόν. Έξι ακροάσεις, κάθε μέρα μία ακρόαση και εμείς λοιπόν είμαστε αρμόδια ή συναρμόδια επιτροπή. Ως επιτροπή λοιπόν εμείς είμαστε υπεύθυνοι για τα επιστολές αξιολόγησης σε έξι ακροάσεις, έξι περιπτώσεις. Είναι τεράστιος ο όγκος δουλειάς για τις επόμενες δέκα ημέρες. Επιπροσθέτως, σε τρεις ακροάσεις πάρα πολύ σημαντικές είμαστε συνεδεμένοι η Επιτροπή, όπως για παράδειγμα για θέματα διαστήματος, ψηφιακή αγορά. Είμαστε συνεργαζόμενοι, συνδεδεμένοι η Επιτροπή για θέματα που αφορούν στην διαστημική πολιτική. Παράδειγμα σας δίνω τώρα. Και σε ό,τι αφορά για την ψηφιακή, σε ό,τι αφορά στην ψηφιακή έννοια αγορά. Σε εννέα ακροάσει δηλαδή ουσιαστικά συμμετέχουμε. Σε έξι μέρες εννέα ακροάσει. και αν προσθέσουμε δε και την ακρόαση του κυρίου Τίμερμαντ. Πρώτο αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτο αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Και θα διεξαχθεί στην αίθουσα τη Ολομέλεια η ακρόαση του με όλους τους επικεφαλείς των πολιτικών ομάδων του Κοινοβουλίου. Άρα, συνολικά καταλήγουμε στις 10 ακροάσεις. Έχουμε ευθύνη για 10 ακροάσεις σε 6 ημέρες. Καμία άλλη λοιπόν δραστηριότητα στην Επιτροπή μας. Δεν έχουμε δραστηριότητες όπως ε, στη σημερινή συνεδρίαση. Ευτυχώ όμω είμαστε στην ώρα μα, ε, έχουμε ξεκινήσει εγκαίρω. Μπορούμε λοιπόν ε, να ξεκινήσουμε τη διαδικασία τη ψηφοφορία. Έχετε τι ε, κάρτε ψηφοφορία. Σα παρακαλώ, βάλτε τι κάρτε στα μηχανήματα και ξεκινάμε. Θέμα λοιπόν είναι ο Γενικό Προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το δημοσιονομικό έτο 2015, όλα τα τμήματα. Να σα ενημερώσω ότι οι 26 τροπολογίες που κατατέθηκαν, μάλλον κατατέθηκαν 26 τροπολογίες. Και τώρα λοιπόν ψηφίζουμε και σε ό,τι αφορά τις συζητήσεις που έγιναν μεταξύ σχεδόν εισηγητών. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Την ψηφοφορία συμβιβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 8. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 9. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Η 10. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. εκεί 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Σεμιβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 26. Ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ γιατί τουλάχιστον δύο ψηφοφορίες θα πρέπει να γίνουν ηλεκτρονικά. Δύο, δύο τουλάχιστον, ναι, πολύ λυπάμαι. Έναρξη ψηφοφορίας ηλεκτρονικά παρακαλώ. Δεν φτάνει μία. Όλοι συμφωνούν. Ναι. Πρόεδρε, τι ψηφίζουμε. Πέρα ψηφοφορία. Την 26, 26. Την 26, πρόεδρε, την 26. Ναι, ναι, ναι, την 26. Πρόεδρε. Διαδικαστικό, πρόεδρε, διαδικαστικό. Γιατί δεν κοιτάτε όταν ε, έχουμε αρνητικούς... Γιατί δεν κοιτάτε στις ε, αρνητικές ψήφους. Κοιτάτε τις θετικές ψήφους, αλλά όχι τις αρνητικές. Ενδιαφέρον αυτό. Ναι, κοιτάξτε, λέει ο πρόεδρος, να σας εξηγήσω. Άμα το 94% της αίθουσας έχει ε, υπερψηφίσει, ε, δεν χρειάζεται να βγω το υπόλοιπο το 6%, το υπόλοιπο 6%. Το βλέπω ξεκάθαρα, δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα. Εάν είναι κρίσιμο και οριακό το αποτέλεσμα, ναι, εντάξει, θα περιμένω μέχρι τέλους. Σας αρκεί αυτή η απάντηση. Όχι, όχι, όχι. Μάλιστα, πέρα της ηλεκτρονικής ψηφοφορία. Α, συγγνώμη, περισσεύουν δύο ψήφοι από τους σοσιαλιστές δημοκράτε. δημοκράτες. Ε, ένας από το ΕΛΚ περισσεύει τώρα. Πολύ λυπάμαι. Είναι πάρα πολύ περίπλοκο. Τελευταία φορά που προσπαθώ να κάνω τέτοιο πράγμα. τη ψηφοφορίας, λοιπόν. Για την 26 ψηφίσαμε και τώρα η ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σύνολο της γνωμοδότησης. Έναρξη της ψηφοφορίας παρακαλώ. Πέρασε. Το αποτέλεσμα είναι μάλλον καλό. 50 ψήφοι υπέρ. Πέντε κατά και μία αποχή. Σας ευχαριστώ πολύ. Πέρας. Now we go to the point number... Και τώρα περνάμε στο σημείο υπαριθμό 9 και 10. Από κοινού θα τα κοιτάξουμε προτάσεις για νομοθεσία σε ό,τι αφορά την ποιότητα της ατμόσφαιρας και τις βιομηχανικές εκπομπές. Πολύ σημαντικές. Δύο προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχουμε παρουσιάσεις της κυρίας Μαρία Βένι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία Μαριάν Βένιν. Α, δεν έχει ακόμα καταφτάσει. Well, we should vote everything electronically because έπρεπε να τα έχουμε ψηφίσει όλα ηλεκτρονικά γιατί να τώρα που τελειώσαμε πιο νωρί και τι πάθαμε. Δεν έχει ακόμα καταφτάσει η αντιπρόσωπο της Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Άρα να περιμένουμε λίγα λεπτάκια. Εμείς στέμε. Που ήμασταν τόσο καλά οργανωμένοι. Ladies and gentlemen. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε. Νομοθετικές προτάσεις για το καθαρό αέρα, για την ποιότητα του αέρα και τις ε, βιομηχανικές εκπομπές. Δύο σημεία, σημείο 9, ε, μείωση εκπομπών κάποιων ατμοσφαιρικών ρήπων που τροποποιεί τον 2003 3-5 και 2035 και περιορισμός εκπομπών ορισμένων ρήπων στην ατμόσφαιρα από μεσαίο γήθους, μεγέθους μονάδες καύσης. Και τα δύο είναι πάρα πολύ σημαντικά, πολύ σημαντικοί κανονισμοί και θα γίνει παρουσίαση από την κυρία Μαριάννε Βένιγκ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. και θα ήθελα να σας ζητήσω ε, να κάνετε μια παρουσίαση 15 λεπτών, ε, μιας και είναι δύο τα θέματα και μετά να γίνει η συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους. Δεν είμαι ο Τόμα Βερχάιρ, όπως σας είπε και ο Πρόεδρος. Ε, είμαι η Διευθύντρια της ε, Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος για την ποιότητα του ζωή και των υδάτων. Και θα σας παρουσιάσω το πρόγραμμα καθαρό Αέρας και ε, τη σχετική νομοθεσία και έγγραφα τα οποία προτείνουμε. Να σας πω καταρχάς ότι η ποιότητα του αέρα ανέκαθεν αποτελούσε σημαντικό ζήτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζετε ότι στη δεκαετία του 70 υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη ατμοσφαιρική ρήπανση και τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να προτείνει νομοθεσία, να εφαρμόσει νομοθεσία και η ατμοσφαιρική ρήπανση βελτιώθηκε, μειώθηκαν οι εκπομπές και θα σας το δείξω αυτό σε ένα λεπτάκι με περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά εξακολουθούμε να δίνουμε μάχη και στο 7ο πρόγραμμα δράσης ε, για το περιβάλλον ε, μας ζητήθηκε να επιτύχουμε ε, στοιχεία ποιότητας τα οποία να μην έχουν πολύ σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις και κινδύνους για την υγεία, την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Αυτό θα πρέπει να το έχετε πάντα κατά νου. Έχετε εδώ αυτή τη διαφάνεια και στην αριστερή πλευρά στο διάγραμμα βλέπετε ότι από το 1990 μέχρι και το 2010 επετέχθη μεγάλη πρόοδος ε, κυρίως ε, σε κάποιους ε, ρήπαντες, τους λεγόμενους σόξ, τους θιούχους, το μονοξίδιο του άνθρακα και τις εκπομπές οξυδιών του αζότου. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι ρηπαντές για τους οποίους έγινε λιγότερη πρόοδος και αυτά είναι τα, ορώματα, τα σωματίδια κυρίως. Και αν δείτε την αριστερή πλευρά της ε, διαφάνειας, βλέπετε και κάποιες ε, ε, καλές εξελίξεις. Έχουμε αποσυνδέσει την ανάπτυξη από την ατμοσφαιρική ρύθμιση, που σημαίνει ότι μπορούμε να έχουμε οικονομική ανάπτυξη χωρίς να έχουμε ατμοσφαιρική ρήπανση. Και αυτό φυσικά είναι ένα πολύ καλό σημείο κίνηση. Παρά την πρόοδο, εκκρεμούν βέβαια κάποια προβλήματα στην Ευρώπη, και να σας δείξω, ε, δείξω τη διαφάνεια, διότι εδώ βλέπετε πόσο σημαντικό είναι το πρόβλημα και το γεγονός ότι εξακολουθεί να υφίσταται. Όσον αφορά την υγεία, για τα αιρούμενα σωματίδια έχουμε ένα πρωτοδιάγραμμα, έχουμε το οξύδιο του, διοξίδιο του αζότου και το όζον. Το όζον ε, ξέρετε ότι είναι οξύδιο του αζότου και πάλι, το οποίο διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο και όλες οι μαύρες κουκίδες που βλέπετε ε, αποδεικνύουν ότι εξακολουθεί να έχει, υπάρχει πρόβλημα ε, με δύο από τους τρεις ρηπαντές και το όζον που δημιουργείται. Και θα θυμάστε βέβαια ότι υπήρχαν και τα τελευταία χρόνια σε διάφορες χώρες και στο Βέλγιο ε, σημεία στα οποία υπήρξε υπερβολική ρήπανση από το λόγο του όζοντος. Και ε, στην τελευταία διαφάνεια έχετε τις παρεμβαλλοντικές επιπτώσεις, τον ευστροφισμό και πολύ μεγάλες ε, εκτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακόμα πλήττονται από ευστροφισμό. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόσκομα. Το πρόσκομα είναι ότι αυτή τη στιγμή η νομοθεσία μας ε, ε, προβλέπει ότι θα πρέπει να επιτύχουμε τις οριακές τιμές για την ποιότητα του αέρα μέχρι το 2015. Αυτό φυσικά είναι αδύνατο και στο πρόγραμμα Καθαρός Αέρας ε, λέμε ότι πρέπει να γίνει μια προσπάθεια να επιτευχθούν οι οριακές τιμές το αργότερο μέχρι το 2020. Και το ερώτημα είναι τι πρέπει να γίνει προκειμένου να φτάσουμε στο στόχο μέχρι το 2020. Από την ανάλυση μας προέκυψε ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία ε, είναι περιορισμένα σε κάποιες γεωγραφικές εκτόσεις και, ε, ε, εκτάσεις και οι τοπικές και περιφερειακές αρχές θα πρέπει να βρουν κατάλληλες λύσεις για να τα αντιμετωπίσουν. Παραδείγματο χάρη σε αστικά κέντρα, στις πόλεις. Αυτό δεν μπορεί να γίνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα ήταν και λογικό να υπάρχει ε, πανευρωπαϊκή νομοθεσία για αυτά. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και το οποίο θα πρέπει να επιλύσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτό είναι το γεγονός ότι ε, δημιουργείται πρόβλημα από τα αυτοκίνητα, από ε, χρήση ε, diesel σε επιβατικά οχήματα. Δείτε εδώ στην δεξιά πλευρά έχουμε το διάγραμμα για τον diesel και βλέπετε ποιες θα πρέπει να είναι οι επιτρεπόμενες τιμές και τι στόχους έχουμε για τη μείωση των εκπομπών και βλέπουμε ότι στο Euro 3 και στο Euro 4 μικραίνει το κόκκινο συννεφάκι. Και αυτό ε, φυσικά μας οδήγησε στο συμπέρασμα ότι η μείωση αυτών των εκπομπών θα ε, είναι εμφανής και στον πραγματικό κόσμο αλλά δυστυχώς βλέπουμε σήμερα ότι οι πραγματικές εκπομπές είναι πολύ υψηλότερε για διάφορους λόγους, δεν μειώνονται και αυτή τη στιγμή είναι τρεις με πέντε φορές πολλαπλάσιες αυτού που θα έπρεπε να είναι. Και αυτό είναι το πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άρχισε ήδη να το αντιμετωπίζει ε, εξετάζοντας τον αναθεωρημένο κύκλο δοκιμών ε, για την έγκριση τύπων ε, συγκεκριμένων οχημάτων και εφαρμόζεται και συγκεκριμένη νομοθεσία μέσω εφαρμοστικών πράξεων θα εφαρμοστεί μέχρι το τέλος του έτους και έτσι θα μπορέσουμε να ε, συμμορφωθούμε με τις τιμές του Euro 6 που θα, θα ξεκινήσουν να ισχύουν από Σεπτέμβριο φέτος και θα μας βοηθήσουν να επιτύχουμε και τους στόχους του 2020 αλλά είναι απορρίτως απαραίτητη και έχει σημασία να ε, θεσπιστεί η συγκεκριμένη νομοθεσία μέχρι το τέλος του έτους. Αυτά λοιπόν για τους στόχους του 2020. Αυτή είναι κείμενη νομοθεσία, την οποία όμως πρέπει να εφαρμόσουμε καταλήλως. Γιατί όμως είναι πρόβλημα η ατμοσφαιρική ρήπανση. Νομίζω ότι οι περισσότεροι από εσά γνωρίζετε ότι σχετίζεται με κίνδυνους για, για την υγεία, καρδιακά προβλήματα, βροχίτιδα και πολλά άλλα. Αλλά θα ήθελα εδώ να σας δείξω και ε, με στοιχεία πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα, διότι ε, τα αιρούμενα σωματίδια και το όζον για παράδειγμα, ε, προκαλούν πρόωρους θανάτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση της τάξης των 406.000 θανάτων το 2010 και φυσικά υπάρχουν και φαινόμενα ευτροφισμού τα οποία ε, πλήττουν κάποιες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτές πλέον αποτελούν το 62%. Οι πρόοροι θάνατοι είναι δεκαπλάσιοι των θανάτων που έχουμε από τροχαία δυστυχήματα. Επομένως δεν είναι ασήμαντο το πρόβλημα και σίγουρα πρέπει να γίνει κάτι. Αν δείτε και την κλίμακα, ε, το χρονοδιάγραμμα μέχρι το 2020, με τα μέτρα τα οποία εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν πολλές, πολύ μεγάλες αλλαγές, υπάρχουν μεν κάποιες μειώσεις οι οποίες δεν είναι ουσιαστικές. Εδώ έχουμε και το κόστος, το οποίο υπολογίζεται ε, σε διάφορα επίπεδα. Έχουμε λοιπόν ένα φάσμα κόστους, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε απόλυτη ακρίβεια εδώ, και βλέπουμε ότι ε, η μονάδα, η τάξη μεγέθους είναι δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο και ε, αυτό αποτελεί το 3 με 9% του ΑΕΠ. Ας δούμε τώρα τι επιτολογές έχουμε από πλευράς πολιτικής για να επιτύχουμε τους στόχους του 2020. Αυτό είναι το πρώτο βήμα πλήρης εφαρμογή των κείμενων μέτρων που διαθέτουμε. Είτε σχετίζονται με εκπομπές, ε, είτε με βιομηχανικές εκπομπές, ε, ε, θιούχα, περιεκτικότητα θείου σε θαλάσσια καύσιμα. Όλα αυτά πρέπει να εφαρμοστούν για να επιτύχουμε το στόχο του 2020 και το πιο σημαντικό είναι οι εκπομπές ρήπων των οχημάτων, των επιβατικών οχημάτων που πρέπει να περάσουν στο Euro 6. Αναφέρθηκα επίσης στην ε, εθνική και τοπική ε, δράση για εφαρμογή από τα κράτη-μέλη. Αυτά μπορεί να τα υποστηρίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των ε, προγραμμάτων LIFE ή οποιοδήποτε άλλων ευρωπαϊκών ταμείων, διαρθρωτικά ταμεία και ούτω καθεξής. Και επίσης πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι η ρήπανση που προέρχεται από άλλες περιοχές, από την Κεντρική Ασία, από τον Κάφκασο, από τη Ρωσία, θα πρέπει να μειωθεί και αυτή, διότι έτσι μειώνεται η διαμεθοριακή ε, ατμοσφαιρική ρήπανση. Υπάρχει το πρότοκολλο του Γκέτεμπερκ, το οποίο το προβλέπει αυτό, αλλά θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι γειτονικέ χώρες ε, θα επιτύχουν τους στόχους και θα πρέπει να τις βοηθήσουμε για τις μειώσεις. Και επίσης ε, θέλουμε να έχουμε και έρευνα και καινοτομία στα πλαίσια του ορίζοντα 2020 πλέον, ώστε να εξεύρουμε νέες λύσεις. Με τους στόχους λοιπόν και τα επιτέγματα του 2020 και τις τιμές της ποιότητας ε, ε, του αέρα, μπορεί να θεωρήσετε ότι το διαχειριζόμαστε το πρόβλημα και θα εξαφανιστεί. Αλλά δεν ισχύει κάτι τέτοιο και θα δείτε εδώ στη διαφάνεια γιατί. Στα αριστερά βλέπετε ότι παρά το γεγονός ότι τηρούνται τα ευρωπαϊκά όρια για την ποιότητα του αέρα και οι οριακές τιμές, για συγκεκριμένα σωματιδία υπάρχει πολύ μεγάλο τμήμα του πληθυσμού που είναι εκτεθειμένο σε ατμοσφαιρική ρήπαση. Είναι λιγότερο για το όζον και είναι πολύ λιγότερο για το διοξίδιο του αζότου, του, ναι, του αλλά νομίζω ότι σε διεθνή βήματα, όπως για παράδειγμα στον ε, ΠΟΕ και στον ΟΣΑ, ε, γνωρίζουν όλοι ότι η ατμοσφαιρική ρήπανση είναι καρκινογόνος πρώτης κατηγορίας και υπάρχουν και κατευθυντήριες γραμμές ε, του ε, ΠΟΗ ε, για τις οριακές τιμές και αν εξετάσουμε εκεί πόσοι άνθρωποι είναι εκτεθειμένοι σε κάποια σωματίδια, παραδείγματο χάρη στο όζον, βλέπουμε ότι έχουμε έκθεση της τάξης των 98% του πληθυσμού που ακόμα εκτίθεται σε ατμοσφαιρική ρήπανση με τις συνέπειες που σας ανέφερα. Πρέπει να προχωρήσουμε λοιπόν παρακάτω και προσπαθούμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε τους στόχους που θα πρέπει να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε για το 2030. Είναι λίγο δύσκολο αυτό το διάγραμμα, αλλά να σας ε, πω δύο λόγια για το τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε. Όσο εφαλτήριο έχουμε το 2005. Βλέπετε ότι Συγγνώμη. Λοιπόν, έχουμε μια μείωση, αυτή είναι η τάση που σας έδειξα προηγουμένως. Αν δείτε την πλέ γραμμή, έχουμε την βασική μείωση. Αυτό είναι αυτό το οποίο θα επιτύχουμε αν εφαρμόσουμε όλα τα μέτρα τα οποία έχουμε ήδη ενεξελίξει και που έχουμε ήδη εφαρμόσει. Μετά έχετε μία ε, κόκκινη, γραμμή και εδώ είναι η περίπτωση στην οποία χρησιμοποιούμε τη μέγιστη τεχνικώς εφικτή μείωση. Είναι όλα τα τεχνικά μέτρα λοιπόν τα οποία έχουμε ήδη ενεξελίξει ε, και είναι καθοδόν και πρέπει τώρα να βρούμε ένα τρόπο να μειώσουμε ε, τις εκπομπές μας με αποτελεσματικό κόστος μεταξύ του κενού αυτού, μεταξύ της βασικής μείωσης που θα έχουμε και της μέγιστης δυνατής. Και εδώ ε, εφαρμόσαμε τα μοντέλα μας, κάναμε κάποιους υπολογισμούς και καταλήξαμε σε ένα σημείο το οποίο θα είναι αποδοτικό προς το κόστος, το οποίο θα μειώσει κατά 52% τις εκπομπές. Εδώ βλέπετε λοιπόν αυτό το 52% ε, το οποίο προέκυψε γιατί στις συζητήσεις που κάναμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν κάνουμε την πρόταση αποφασίσαμε να φύγουμε λίγο από το πιο αποτελεσματικό το κόστος σημείο, ε, διότι διαπιστώσαμε ότι σε κάποιους τομείς, ε, στη γεωργία, ε, για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να μειώσουμε το κόστος αποτελεσματικά χωρίς να χάσουμε τα ωφέλη. Εδώ λοιπόν φτάνουμε σε αυτό το μείον 52% και εδώ έχουμε την πράσινη γραμμή που έχει και αυτή τη σημασία της, διότι εδώ έχουμε συνδυάσει το μοντέλο για την ποιότητα του αέρα με τα όσα συμβαίνουν ε, στην, ε, στο θεματολόγιο της κλιματικής αλλαγής. Ε, έχουμε και το πρόγραμμα για την ενέργεια για το 2030, το οποίο θα έχει θετικές συνέπειες για την συμβατική ατμοσφαιρική ρήπανση και αν τεθεί σε εφαρμογή αυτή η δέσμη μέτρων, και αυτό ακόμα εκρεμεί, θα μπορούσαμε να φτάσουμε στο μείον 65%. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό λοιπόν και θα πρέπει να το έχουμε κατά νου. Οι προτιμόμενες λοιπόν επιλογές πολιτικές, ε, πολιτικής για το 2030 είναι ότι με τις πολιτικές τις οποίες θα σας δείξω ε, σε ένα λεπτό μπορούμε να μειώσουμε τις συνέπειες για την υγεία κατά 52% την επιφάνεια η οποία πλήττεται από ευστροφισμό κατά 35% και την οξύνηση ε, κατά 85%. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε μείωση εκπομπών των 6 βασικών ρηπαντών μέχρι το 2020 ε, και το 2030 στη συνέχεια, δεν θα σας δώσω όλα τα αριθματικά στοιχεία γιατί δεν υπάρχει λόγος, αλλά τα στοιχεία τα οποία έχουμε εδώ είναι αυτά τα οποία θα θέλαμε να επιτύχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην νομοθεσία έχουμε κάνει διαφοροποίηση για κάθε ένα ε, κράτος μέλος. Υπάρχουν ευελιξίες, διότι κάποιοι από τους στόχους ε, είναι φιλόδοξοι, μπορώ να το πω αυτό, αλλά υπάρχουν και κάποιοι μηχανισμοί εκκίνησης, ε, ε, βάσει των οποίων, για παράδειγμα, θα μπορούσαν να μειωθούν τα κάψιμα στη θάλασσα. Επίσης, έχουμε και κάποια στοιχεία όταν διαπιστώνουμε ότι έχουμε ανακαλύψει κάτι καλύτερο στα, στα αρχεία μας. Ε, τα βασικά στοιχεία του προγράμματος τα γνωρίζετε, δεν θα σας τα διατράξω αυτά. Περνάω κατευθείαν στην ε, αναθεώρηση της οδηγίας για τις ε, δεσμεύσεις για τις εθνικές εκπομπές ατμοσφαιρικών ρήπων και μετά θα περάσω στις μεσαίου μεγέθους μειονάδες καύσεως. Λοιπόν, για τις εθνικές εκπομπές είπαμε ότι έχουμε έξι βασικά ρηπαντές και από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφορα στάδια μέχρι το 2020. Ε, στο 2020 είναι το πρωτόκολλο του Γκέτεμπορκ, είναι κάτι το οποίο έχει ήδη συμφωνηθεί, διότι αποφασίστηκε ε, το τέλος του 2012 στο Γκέτεμπορκ. Κατόπιν, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι από το 2020 στο 2030 θα τηρήσουμε την πορεία που έχουμε προβλέψει, έχουμε βάλει ένα ενδιάμεσο σημείο ελέγχου το 2025, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι τα κράτη-μέλη ε, δεν θα ξεκινήσουν καθυστερημένα. Το πρόβλημα που έχουμε τώρα με την νομοθεσία μας και ε, ο λόγος για τον οποίο δεν μπορούμε να επιτύχουμε τις συγκεκριμένες οριακές τιμές είναι γιατί τα κράτη-μέλη ξεκίνησαν λίγο καθυστερημένα. Είναι δύο, καταλαβαίνετε. Μάλιστα. Σας μίλησα λοιπόν για τα άλλα σημεία σε ό,τι αφορά την πρόταση για τις, για τις ε, ε, εργοστάσια καύσης. Είχαμε λοιπόν την οδηγία για το οτιδήποτε που ήταν ε, κάτω από 10 ΜΒ και ύστερα και την άλλη οδηγία για πάνω από το όριο αυτό. Τρεις ρηπαντέ ε, ε, ρηπαντές είχαμε σε ό,τι αφορά τον OXPM. 20% της μείωσης μπορούμε να την πετύχουμε μέσω των μέτρων αυτών και ήμασταν πάρα πολύ επιλεκτικοί. Κοιτάξαμε τα μεμονωμένα σημεία σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, σε ό,τι αφορά τους καυστήρες, τις ε, τουρμπίνες και άλλα είδη εργοστασίων, υφιστάμενα εργοστάσια και νέα εργοστάσια. Έχουμε λοιπόν μεγάλη ευελιξία και ανάλογα ε, έχουμε οργανώσει και την εφαρμογή. Θα τα κοιτάξουμε λίγο παρακάτω αυτά. Το διοικητικό άκτο το κρατήσαμε αρκετά χαμηλό γιατί δεν ε, ζητήσαμε αδειοδότηση αλλά καταγραφή μόνο. Τελευταία διαφάνεια, κύριε Πρόεδρε. Έχουμε λοιπόν συγκεκριμένα ωφέλη και συγκεκριμένα, συγκεκριμένα κόστος για το 2030. Βλέπουμε ότι η μείωση του εξωτερικού κόστους μπορεί να είναι μεταξύ 44 και 140 δισεκατομμυρίων ευρώ ανά έτος και αυτό περιλαμβάνει ε, την εξοικονόμηση άμεσου κόστους, 3 ε, δισεκατομμύρια δηλαδή σε ό,τι αφορά ε, το υγειονομικό κόστος που εξοικονομείται σε ό,τι αφορά το κόστος ε, εφαρμογής από την άλλη. Είναι ουσιαστικά λίγο πολύ το ίδιο όπως και το άμεσο κόστος το οποίο εξοικονομείται, 3,3 δισεκατομμύρια ανά έτος. Αλλά και αυτό μπορεί να καταστεί πιο φθηνό εάν το πακέτο για το κλίμα και την ενέργεια το 2030 εφαρμοστεί. Έχουμε λοιπόν συνολικό θετικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη του ΑΕΠ και στην αναπασχόληση, περίπου 12 έως 40 φορές χαμηλότερο το κόστο από ό,τι τα ωφέλη. λοιπόν ότι είναι πολύ ισορροπημένο το πακέτο αυτό. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσοχή σα. Σα ευχαριστούμε. Κυρία Βένιγκ. Θα έχουμε την ευκαιρία στη διάρκεια των απαντήσεων να αναπτύξουμε πιο διεξοδικά το θέμα το δεύτερο, γιατί περισσότερο επικεντρωθήκατε στο πρώτο. Το πρώτο είναι πιο γενικό και το δεύτερο είναι πιο ειδικό για τις μεσαίες μονάδες καύσης. Εμείς έχουμε δύο γνωμοδοτήσεις και δύο συντάκτες γνωμοδότησης. Για την πρώτη οδηγία την μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρήπων, με τροποποίηση της οδηγίας 35 του 2003, συντάκτης του γνωμοδότης είναι ο κύριος Γκέρεκ από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Παρακαλώ κύριε Γκέρεκ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα περιοριστώ στο περιεχόμενο της οδηγίας γιατί η κυρία Διευθύντρια μίλησε για, σωστά για κάποια γενικά θέματα, αλλά εγώ θα ήθελα να επανέλθουμε στα συγκεκριμένα θέματα, στο ίδια, στην ίδια την οδηγία. Η προτινόμενη οδηγία λοιπόν αποτελεί συνδυασμό μερικών ε, προηγούμενων ε, κειμένων, την οδηγία του 2001, την οδηγία του 2003, του πρωτοκόλου του Γκέτεμπορκ του 1999, των ανακοινώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόκειται για μια συμπίληση κειμένων ουσιαστικά. Ο στόχος της νέας οδηγίας, αυτό αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο νέο της σχέδιο, της 18ης Δεκεμβρίου του 2013 για, για τον περιορισμό εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρήπων. Στόχος λοιπόν είναι η ενίσχυση της καινοτομία ε, και της οικολογικής ανάπτυξης της οικονομίας, της, της ε, ανταγωνιστικότητας, την προστασία των φυσικών πόρων και τη δημιουργία οικολογικών τεχνολογιών. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν μιλούμε για ένα συνδυασμό, για μια συμπίληση νομοθετικών κειμένων. Ποιο είναι το καινούριο στοιχείο της, του νέου σχεδίου της οδηγίας. Αυτή είναι η ερώτησή μου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι το καινούριο προσφέρει η νέα οδηγία. Έχω και κάποιες παρατηρήσεις ε, για την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρώτον, ε, στο σχέδιο δεν, υπό, δεν υπόψη όλες, ε, όλα τα, όλες οι εκπομπές, κυρίως των αιωρούμενων σωματιδίων που έχουν διάμετρο μικρότερη από τα 2,5 εκατομμύρια στάτου μέτρου. Τα σωματιδία είναι τα πιο επικίνδυνα και για την υγεία και για το κλίμα, γιατί έχουν νανομετρικά μεγέθη αυτά τα αιωρούμενα σωματίδια. Επίσης δεν λαμβάνονται υπόψη χλωριωμένοι αρωματικοί υδρογονάνθρακες, δηλαδή διοξίνες. Επίσης παραλείπονται συγκεκριμένες ε, εποχιακές εκπομπές, την εποχή της θέρμασης, οι χαμηλές εκπομπές για παράδειγμα, ούτε αυτές έλειψαν υπόψη. Είναι σημαντικό αυτό το θέμα, κυρίως για την τοπική αυτοδιοίκηση. Θα πρέπει όμως και εδώ να δώσουμε κάποια ενάυσματα και να έχουμε μια νομοθετική ρύθμιση. Χαμηλέ χαμηλές πολύ σημαντικό. Επίσης, παραλείπονται κάποια επικίνδυνα αέρια που εκλείονται σε μεγάλες ποσότητες και είναι ανθρωπογενικής προέλευση, όπως το υδρόθιο για παράδειγμα. Επίσης θα ήθελα πιο διεξοδική ανάλυση της ευελιξία που υπάρχει στην καταμέτρηση των εκπομπών. Περί τίνος πρόκειται. Μήπως έχουμε εδώ κάποια τεχνάσματα, κάποιους συνδυασμούς για κάπως παραποιημένη καταμέτρηση. Και έχω και μία μορφή για το τυπικό της οδηγίας. Για παράδειγμα, παραπέμπει η οδηγία σε διαφορετικά παραρτήματα που είναι διάσπαρτα σε άλλες νομοθετικές πράξεις. Αυτό δημιουργεί χάος και αδιαφάνεια στο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θεωρώ ότι η πρόταση οδηγίας θα πρέπει να έχει τα δικά της παραρτήματα και να μην παραπέμπει αριστερά και δεξιά σε διάφορα άλλα παραρτήματα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Σίγουρα υπάρχουν θετικά στοιχεία στην οδηγία. Ε, παρακαλώ, λάβετε υπόψη και σημειώστε και τα σχόλια του συναδέλφου για να μπορέσετε να απαντήσετε αργότερα. Και τώρα θα ακούσουμε τη, το συντάκτη της Γνωμοδότηση για το δεύτερο θέμα, τον περιορισμό των εκπομπών ορισμένων ρήμων στην ατμόσφαιρα από μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης. Συντάκτης γνωμοδότησης είναι ο κύριος Φέντερλεϊ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Οι δύο οδηγίες είναι πολύ σημαντικές και για το κλίμα και για το περιβάλλον και για την υγεία αλλά και για την οικονομία. 4.000 ε, ε, πρόωροι θάνατοι λέμε ότι κατά πάσα πιθανότητα οφείλονται σε αυτή την ατμοσφαιρική ρήπανση με κόστος ε, μεταξύ 300 δισεκατομμύριων και 940 δισεκατομμύριων ευρώ κόστος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλά χρήματα λοιπόν φεύγουν από τις τσέπες των φορολογουμένων για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και για να μην μιλήσουμε για τους πρόωρους θανάτους. Μιλάμε για μεγάλες ψηφίδες ενός ευρύτερου ψηφιδωτού που αφορά το περιβάλλον και γεμίζει το κενό μεταξύ της οδηγίας για, τα, ε, ε, για τις μεσαία μεγέθους μονάδες καύσης και της, ε, την οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές. Έχουμε 143.000, επαναλαμβάνω 143.000 χιλιάδες, 143 ε, εκατομμύρια μάλλον ε, μεσαίου μονάδος καύσης για θέρμανση, ε, παραγωγή ηλεκτρισμού, παροχή ζεστού νερού και ψήξη. Έχουμε τεράστια κατανάλωση. Λοιπόν, οι περισσότερες μονάδες καύσης είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οπότε θα πρέπει να φροντίσουμε η γραφειοκρατία των ε, νέων ε, νομοθετικών ρυθμίσεων να μην επιβαρύνει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης ε, θα θέλαμε εξασφάλιση συνθηκών ίσου ανταγωνισμού. Ιδιαίτερα να μην επιβαρύνουμε την δημοτική θέρμανση, επιχειρήση δημοτικής θέρμασης, μικρής εμβέλειας. Επίσης θέλουμε η νέα νομοθετική την ρυθμίση να εντάσσεται στις περιβαλλοντικές ρυθμίσεις και να συνάδουν με την περιβαλλοντική νομοθεσία ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην βρεθούν σε δυσμενή θέση κάποιες εναλλακτικέ φιλικές προς το περιβάλλον. Οι προτάσεις είναι θετικές για το περιβάλλον. Θα μας εξασφαλίσουν και ασφαλέστερη ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά θα μας εξοικονομήσουν και τεράστια ποσά από τη στιγμή που θα εφαρμοστούν οι νέες ρυθμίσεις. Σας ευχαριστώ. Και τώρα να σας ζητήσω ε, να δώσουμε το λόγο στους κοιόδες εισηγητής για την οδηγία για τα εθνικά για τα, όρια των εθνικών επιτροπών η κυρία Γελκούνεν από το ΕΛΚΑ έχει το λόγο Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εξαιρετική της ε, παρουσίαση. Το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το πακέτο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για, την, ε, το περιβάλλον. Είναι εξαιρετική η στοχοθεσία. Παρ' όλα αυτά, το θέμα τώρα είναι πώς θα τεθούν πιο δεσμευτικοί και φιλόδοξοι στόχοι. Ξέρετε ποιες ήταν οι συνέπειες, ποιες ήταν αντίκτυπος της τρέχουσας οδηγίας και πόσο αξιόπιστες είναι οι πληροφορίε, τα δεδομένα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας. Από την άλλη ακούμε ότι με τι διάφορε οδηγίε. κοιτάμε και την ίδια τη βιομηχανία και πιστεύουμε ότι αυτή η προσέγγιση, αυτή η νέα προσέγγιση θα έχει επιπτώσεις και στον αγροτικό τομέα. σε ό,τι αφορά τις εκπομπές σε μεθανείο κτλ και αμμονίας. Ξέρετε λοιπόν ε, ποιοι τομεί ε, θα αναγκαστούν να φέρουν το κόστος αυτό και αφετέρου πώς θα διαμορφωθεί η ευελιξία στα πλαίσια της οδηγίας αυτής, γιατί ξέρουμε ότι τα γεωγραφικά δεδομένα είναι πολύ διαφορετικά στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλιά σας. Σκύοντας εισηγητής για τις μεσαίες μονάδες καύσης από πλευράς του ΕΛΚ. Ο κύριος Ρόιλ έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, όλα αυτά ακούγονται πολύ καλά και πολύ σημαντικά γιατί φυσικά όλοι θέλουμε να βελτιώσουμε την ατμόσφαιρα και το περιβάλλον. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια να τα κοιτάξουμε όλα αυτά σε επίπεδο μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Το είπε και ο συνάδελφο και αυτό και η συνάδελφο που μίλησε πριν από λίγο. Και υπάρχουν κάποιε ε, υποδείξει τι οποίε θα πρέπει να τι κοιτάξουμε με επικριτικό μάτι. Σε ό,τι αφορά τα όρια τα οποία έχουν ήδη τεθεί, έχουν, ε, είναι, δεν είναι πολύ φιλόδοξα και θέλουμε λοιπόν να μειωθούν. Οι ειδικοί, οι εμπειρογνώμονε του ε, οποίου ρώτησα, μα είπαν ότι δεν είναι πλέον οικονομικά από το δική αυτή η προσέγγιση. Θα πρέπει λοιπόν να το σκεφτούμε αυτό, μήπω θα πρέπει να το σκεφτούμε πρωτού πάρουμε αποφάσει. Και θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώ κατέληξε σε αυτέ τι προτινόμενε οριακέ τιμέ και στην πρόταση μείωση του. Γιατί δεν έλαβε υπόψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα εφιστάμενα εργοστάσια, τι εφιστάμενε μονάδε. Λέμε ότι όλο και πιο πολύ θέλουμε να σκεφτόμαστε ποιε είναι οι συνέπειε των αποφάσεών μα. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να πούμε ότι ως τώρα έχουμε ενδεχομένως κάποιες φιλοδοξίες, κάποια όνειρα, αλλά όχι συγκεκριμένα αντίληψη για το ποιος θα είναι αντίκτυπος. Σε ό,τι αφορά την ετήσια προσμέτρηση, πώς θα γίνουν αυτά, πώς θα γίνει αυτή η ετήσια προσμέτρηση, γιατί βελτιώνεται το σύστημα αυτό. Μήπως πρόκειται για μια απόπειρα να επιβληθεί ένα νέο ε, βραδύ σύστημα. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πολύ γραφειοκρατική αυτή η διαδικασία έκτος και αν μπορείτε να μας εξηγήσετε ποιες είναι οι ε, για την πολιτική. Και το ίδιο σημαίνει και ισχύει και για την τη περίοδο. Μία μικρή παρατήρηση. Μιλάμε για μία δεκαετή υποχρέωση διατήρησης των δεδομένων αυτών. Τι πλέον έχει αυτό το σύστημα. Μήπως απλά γεμίζουμε ντουλάπια. Ποιος είναι, ποιος είναι ο σκοπός του μέτρου αυτού. Πολύ φοβάμαι δηλαδή ότι ε, ρυθμίζουμε και πάλι υπερβολικά πολλές λεπτομέρειες, οι οποίες δεν χρειάζονται να ρυθμιστούν. Μιλάμε για ένα δημόσιο μητρό για τις ε, ε, μεσέ και μεγάλες τέτοιε μονάδε καύση. Γιατί έω τώρα προβλεπόταν μόνο για τι μεγάλε μονάδε καύση. Γιατί τώρα περιλαμβάνονται και μεσέ, για πείτε μου. Και Θεωρώ ότι στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γίνεται η αναφορά ότι κάθε τεχνική παρατήρηση ε, γίνεται οξύδωση και όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται στην οδηγία αυτή. Υπάρχουν όμως μέσα ε, ε, μονάδες που καλύπτονται ήδη από την οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές. είναι επικάλυψη είναι αυτό λοιπόν έξυπνο. Είναι απαραίτητο. Δεν θα πρέπει να υπάρχει μια σαφή μια σαφή δάκρυση. Την επόμενη εβδομάδα, την ε, επόμενη εβδομάδα θα κάνουμε ακρόαση των επιτρόπων και ένα σημαντικό εργαλείο είναι ο πρώτος αντιπρόεδρος ο οποίος θέλει να επιβάλλει καλύτερη νομική βεβαιότητα. Νομίζω ότι αυτό είναι απαραίτητο να το θέσουμε ως έργο. Καλή είναι και η μεγάλη σχόλια, αλλά δεν γίνεται όταν καλούμαστε να αποφασίσουμε τις λεπτομέρειες, να αποφασίσουμε αντίθετα πράγματα. Θα πρέπει λοιπόν κάθε λεπτομερές μέτρο να είναι όπως είναι. Θα πρέπει να υπάρχει προθυμία να κάνουμε και συγκεκριμένες αλλαγές. Και όχι μόνο να χανόμαστε στους μεγάλους στόχους. Ευχαριστώ πάρα πολύ συνάδελφε. Η κυρία Μία Πέτρα Κουμπούλανάτρη είναι σκιώδης συγγήτρια σε ό,τι αφορά τις μεσαίες μονάδες καύσης και έχει το λόγο από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μιλήσω και εγώ φιλανδικά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για την ε, παρουσίαση που μας έκανε. Νομίζω ότι είναι σημαντικός αυτός ο στόχος ε, της βελτίωσης της ποιότητας του αέρα. Το θέμα αφορά και τη βιομηχανία και την ενέργεια άρα εμπίπτει πλήρως στις αρμοδιότητες της Επιτροπής μας. Ο κλάδος της ενέργειας ε, και οι σχετικές επιχειρήσεις θα πρέπει να μειώσουν τις ε, εκπομπές αερίων τους και καλό θα ήταν να αντικαταστήσουν ε, τα καύσιμά τους από βιομάζα σε μεγάλο βαθμό γιατί υπάρχουν πολλές δυνατότητες αντί να έχουμε καύση να χρησιμοποιούμε βιομάζα. Έτσι αποφεύγουμε και το κόστος μεταφοράς ε, των καυσίμων. Θα πρέπει να εξετάσουμε το πρόβλημα και περιφερειακά, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε περιφέρειας, αλλά και την αποφυγή αντιφατικών στόχων. Οι μονάδες καύσης θα πρέπει να είναι μεσαίου μεγέθους οι αποτεθρωτήρες δηλαδή και Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι η συνεχής παρακολούθηση, η συνεχής εποπτεία. Βέβαια αυτό ίσως δημιουργήσει πρόβλημα στις μικρού μεγέθους μονάδες. και η βιομηχανία μπορεί να έχει πρόβλημα, γιατί οι μικρές ε, μονάδες καύσης ε, χρησιμοποιούν καύσιμα από τα απόθεμά τους και εκεί θα πρέπει να δούμε αν μπορούμε να βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας ώστε να βελτιώσουμε και τη δημόσια υγεία. Σίγουρα θα πρέπει να βελτιώσουμε την ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε, αλλά ταυτόχρονα να προωθήσουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η κυρία Μισελ Ριβαζή, που είναι σκιώδη συγγήτρια και για τις δύο προτάσεις εκ μέρους των Πρασίνων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίαση που μας έκανε και που δείχνει ότι όταν έχουμε κείμενα Έχουμε βελτίωση και της ανάπτυξης όπως είπατε, αλλά έχουμε βελτίωση και της υγείας γιατί όταν έχουμε μια οδηγία για την ατμοσφαιρική ρήπανση, στόχος μας είναι να βελτιώσουμε τη δημόσια υγεία. Γιατί το κόστος της υγείας ε, είναι κάθε χρόνο 940 δισεκατομμύρια σε δαπάνες στην υγεία και 400.000 άνθρωποι χάνουν πρόωρα τη ζωή τους. Για να μην αναφέρω το πρόβλημα του ευτροφισμού σημαντικά, σημαντικές προκλήσεις λοιπόν και κυβεύματα και ε, αν προσθέσουμε και το μεθάνιο στη νέα οδηγία έχουμε και μία επίπτωση στα αέρια του θερμοκηπίου. Άρα έχουμε και περιβαλλοντική ε, πολιτική. Έχουμε 21% πιο επιβαρυντικά από το διοξείδιο του άνθρακα. Και ε, ε, τι γίνεται με τα αιρούμενα σωματίδια διαμέτρου 2,5 εκατομμυριωστών, γιατί αναφέρεται μόνο τα 10. Γιατί δεν, περιλαμβάνετε, δεν περιλάβατε και τον υδράργυρο. Εμείς ζητήσαμε και ο υδράργυρος να περιληφθεί στη νέα οδηγία, γιατί είναι ενδοκρινολογικός διαταράκτης ο υδράργυρος. Επίσης διαπιστώνουμε ότι πάνω από 20 χώρες δεν σέβονται τους κανόνες ξεκίνησε μια διαδικασία επιβολή κυρώσεων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει να δώσουμε περισσότερα ενάψματα, γιατί η βιομηχανία έκανε το καθήκον της, αλλά στις πόλεις έχουμε πληθώρα προβλημάτων εξαιτίας των εθνικών πολιτικών που μένουν α, α, αριθμιστά. Και αναφέρατε την περίπτωση του ντίζελ. Μας δώσατε τον πίνακα για τους στόχους του 2030. Γιατί δεν ευθυγραμμιστήκατε για τους στόχους αυτούς ε, με, του, με τους στόχους ε, του σχεδίου για το κλίμα με μείωση κατά 40% των ε, καυσαερίων, των αερίων του θερμοκηπίου, θα μπορούσατε να είστε πολύ πιο φιλόδοξοι στην πρότασή σας. Γιατί δεν το κάνατε. Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη οδηγία τώρα, για τις μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης. Το θέμα εδώ είναι επίγον. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, έχουμε πολλά εργοστάσια, πολλές μονάδες που χρησιμοποιούν τη βιομάζα και εντάσσονται πλήρως στην οδηγία, γιατί μέχρι στιγμής δεν είχαμε κανόνες για τις περιπτώσεις αυτές. Χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερως για την πρόταση οδηγία σας, γιατί ε, τα εργοστάσια της βιομάζας που θα καλύπτουν πάνω από 900.000 τόνους ξύλου στην Καρτάν, μια ε, περιοχή με μεγάλη ατμοσφαιρική ρήπανση και χαιρόμαστε που υπάρχουν αυτά τα νέα μέτρα και αυτό θα πρέπει είτε να ε, επιβάλλουμε δρακόντια μέτρα για να περιορίσουμε αυτές ε, τις μονάδες που χρησιμοποιούν βιομάζα γιατί επιβαρύνουν ε, το περιβάλλον και ελπίζω να μειώσουμε αυτά τα μεγάλα εργοστάσια που υπό το πρόσχημα ε, της, ε, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ε, επιβαρύνουν και την ατμόσφαιρα με πολλούς ρήπους αλλά και αποψηλώνουν τα δάση με την καύση τεραστιών ποσοτήτων ξυλίας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Άσλι Φόξ είναι ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ομάδα των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών συμμερίζεται την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι πρέπει να βελτιώσουμε την ποιότητα του αέρα, αλλά μας υπενθυμίζουν πάντα τι συνέπειες έχουν οι καλές προθέσεις και χαίρομαι που ο κύριος Ρόιλ συνεισέφερε στη συζήτηση. Συμφωνώ με πολλά από αυτά τα οποία μας είπε σήμερα. Δεν υπάρχει νόημα να επιβάλλουμε ακόμα αυστηρότερο περιβαλλοντικά όρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν αποτέλεσμα οι βιομηχανίες μετεγκαθιστούνται εκτός Ευρωπαϊκής, μετεγκαθίστανται Ευρωπαϊκής Ένωσης και παράγουν το ίδιο προϊόν, προϊόν κάπου αλλού, εκπέμποντας πολύ περισσότερες ε, ρηπογόνες ουσίες στην ατμόσφαιρα και εμείς ε, στη συνέχεια εισάγουμε αυτά τα προϊόντα στις χώρες μας. Και φοβάμαι ότι αυτή είναι η παρενέργεια κάποιων από τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχει, για παράδειγμα, ένα εργοστάσιο αλουμινίου στη βορειοανατολική Αγγλία που ε, έκλεισε και ε, μετεγκαταστάθηκε στον Καναδά. Είναι κλασικό παράδειγμα ε, του γεγονότος ότι δεν ε, μειώσαμε την ρήπανση που εκπέμπεται στην ατμόσφαιρα, απλώς μεταφέραμε το εργοστάσιο κάπου αλλού. Χρειαζόμαστε κατάλληλο ποσοστό ευελιξίας για τα κράτη-μέλη, ώστε να μπορέσουν να επιτύχουν αυτούς τους στόχους. Ε, υποστηρίζουμε τους στόχους σας λοιπόν Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη βελτίωση του αέρα που αναπνέουμε, αλλά θέλουμε να επιτευχθεί αυτό κατά τρόπον ώστε να προστατευτούν όσο το δυνατόν περισσότερες θέσει εργασία και όσο περισσότερες βιομηχανίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, συνάδελφε. Ήγηκε η ώρα των απαντήσεων και των καταληκτικών σας ε, παρατηρήσεων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ όλους για τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Δεν ε, θα απαντήσω σε ερωτήσεις μία προς μία, ελπίζω να συμφωνείτε. Θα προσπαθήσω να τις ομαδοποιήσω λίγο και ελπίζω να σας δώσω κάποιες ικανοποιητικέ απαντήσεις. Καταρχάς, να σας πω ότι υπήρξαν και κάποια ενθαρρυντικά σχόλια και αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν κάποιες ανησυχίες για κάποια θέματα και είμαστε και μαθημένοι, διότι έγινε μια πολύ μακρά σε προπαρασκευής, ε, τρία-τέσσερα χρόνια διαβουλεύσεις με τους ενδιαφορομένους, με όποιον μπορείτε να φανταστείτε. Ε, από τον κλάδο, πολύ μεγάλες ε, μονάδες καύσης, ε, γεωργία, μεταπητική βιομηχανία. Δεν θέλω να του αναφέρω έναν προς έναν, αλλά υπήρχε συμμετοχή όλων σε αυτή τη διαδικασία και είχα την ευκαιρία να ακούσω τα σχόλιά του και να συνεργαστώ μαζί τους αν υπήρχαν κάποια θέματα τα οποία με ανησυχούσαν ιδιαίτερα. Δεύτερον, χρησιμοποίησαμε τα πιο προηγμένα μέσα μοντελοποίησης που είχαμε στη διάθεσή μας. Ξέρω ότι η μοντελοποίηση ορισμένες φορές ε, μπορεί να δημιουργήσει ανησυχίες, ε, διότι δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα, αλλά είναι ότι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Δεν μπορούμε να πάμε πέρα από αυτόν, κάπως πρέπει να εμπιστευτούμε αυτό το σύστημα. Επιπλέον, ε, εξετάσαμε και μακροοικονομικές συνέπειες και συνέπειες αυτού του είδους, όχι μόνο περιβαλλοντικές συνέπειες, αλλά και μακροοικονομικές συνέπειες εν γέννη και επιπλέον, επειδή αυτό προέκυψε και από τη συζήτηση, συμπεριλάβαμε και τη δέσμη μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια, τα οποία είναι προς συζήτηση και προσυμφωνία. συμφωνία. Όταν λοιπόν ε, λέτε ότι ίσως θα μπορούσαμε να πάμε ε, λίγο παρακάτω, ναι, θα μπορούσαμε να πάμε λίγο παρακάτω αν εφαρμοζόταν σωστά αυτή η δέσμη μέτρων και αυτό περιλαμβάνεται και ε, στις διαφάνειές μου, ε, σας το έδειξα. Εάν συνδυάσουμε δυνάμεις με το κλίμα και την ενέργεια, ίσως θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Αλλά δεν έχει νόημα να προτείνουμε εμείς μέτρα τα οποία ούτως ή άλλως περιλαμβάνονται αλλού γιατί δεν θα βοηθήσει σε τίποτα. Αυτά λοιπόν επιγραμματικά. Τώρα, ε, κάποιες ερωτήσεις αναφέρθηκαν στις δυσκολίες από πλευράς κόστους ε, για το κατά πόσον ο κλάδος ε, μπορεί να αντέξει αυτό το κόστος. Εμείς εξετάσαμε τις λύσεις οι οποίες είναι οι περισσότερο αποδοτικές ως προς το κόστος. Ε, εάν εξετάσετε τα θέματα θα δείτε ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι και κυρίως ο κλάδος και το κλάδος των αυτοκινήτων οχημάτων έχει κάνει μεγάλη προσπάθεια και στα πλαίσια της συγκεκριμένη ε, νομοθεσίας και αυτό είναι αποδεκτό από όλους, γι' αυτό ακριβώ και δεν προτείνουμε νέα νομοθεσία μέχρι το 2020. Υπάρχουν όμως κάποιοι κλάδοι οι οποίοι όσον αφορά τα μέτρα τα οποία λήφθηκαν για να μειώσουν τις εκπομπές, υστερούν. Παραδείγματος χάρη, ο γεωργικός τομέας δεν έχει κάνει και πάρα πολλά από το 1990 μέχρι σήμερα και αν δείτε την επιλογή που είναι πιο αποτελεσματική ως προς το κόστος, τότε καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι μπορούμε να το μειώσουμε με το χαμηλότερο κόστος και εκεί κυρίως ε, εν μέρη είναι και ο κλάδος της γεωργίας. Υπάρχουν όμως και κάποιοι κλάδοι οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν αναλάβει μεγάλο μερίδιο ευθύνη και προσπαθούμε να μειώσουμε το κόστος και για αυτούς, μειώνοντας τους στόχους μας, ε, τους στόχους που θέλουμε να πετύχουμε και βελτιώνοντας έτσι και το κόστος για τον τομέα της γεωργίας και για κάποιους άλλους βιομηχανικούς κλάδους. Δεν είχαμε αρνητικές απαντήσεις από τον κλάδο όπως έλαβα από κάποιους από εσά εδώ ε, στις προτάσεις μας. Ίσως γιατί μπήκαμε σε μια διαδικασία ε, εκτεταμένης διαβούλευσης. Να σταθώ τώρα σε κάποια συγκεκριμένα θέματα. Νομίζω ότι κάπου για τις μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσεως αναφέρθηκε ότι δεν περιλαμβάνονται ε, τα ε, αιωρούμενα σωματίδια. Ε, όχι, τα έχουμε συμπεριλάβει αυτά. Δεν έχουμε συμπεριλάβει κάποια άλλα αέρια, διότι το ελέγξαμε με τον Μπόι και θεωρήθηκε ότι δεν είναι πολύ μεγάλο ε, το ποσοστό ανησυχίας, επομένως δεν θεωρήθηκε ότι είναι απαραίτητο να ληφθούν και αυτά υπόψη. Κάναμε τους οπολογισμούς της μείωσης, όπως σας είπα, με τρόπο ο οποίος θα είναι πιο αποτελεσματικό αποτελεσματικός και ως προς τη δαπάνη μας και ε, εξετάζουμε και ευελιξίες ε, όσον αφορά τα χρονοδιαγράμματα. Και εδώ να επανέλθω σε κάποια από τα σχόλια που ακούστηκαν ότι ε, ναι γίνεται μετεγκατάσταση. Δεν υπάρχει λόγος μετεγκατάστασης, ιδίω για, τα μεσαίου για τις μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης, που ούτως ή άλλως είναι μικρότερες μονάδες. Τι κάναμε. Έχουμε κάνει μια βαθμιδόν εφαρμογή ε, για τις μικρές μονάδες από 1 έως 5 ΜΒ δεν υπάρχει υποχρέωση εφαρμογής αυτής της νομοθεσίας μέχρι το 2030 για ε, την υφιστάμενη νομοθεσία τώρα. Ε, ο, για οποιαδήποτε νέα νομοθεσία θα πρέπει να υπάρχει συμμόρφωση σχετικά γρήγορα. Αυτή τη στιγμή τεθεί σε ισχύ η νέα νομοθεσία. Αλλά είναι νέε οι μονάδε ούτω ή άλλω, επομένω δεν υπάρχουν τα τεχνικά προβλήματα. Για τι υφιστάμενες μονάδε υπάρχει μια μακρά περίοδο προσαρμογή και ε, η τιμές εκπομπών είναι διαφορετικές για τις μεγαλύτερες και μεσαίες μονάδες. Έχουμε κινητήρες, τουρμπίνες, καυστήρες, όλα αυτά είναι ξεχωριστά, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι λαμβάνονται υπόψη οι ειδικέ συνθήκε που επικρατούν σε κάθε μία από αυτέ τι μονάδε. Όσον αφορά τη βιομάζα τώρα, να σας πω ότι Όντως ήταν πολύ μεγάλο το πρόβλημα, γι' αυτό ακριβώς και εδώ συνδυάσαμε τις δυνάμεις μας με τους συναδέλφους από το κλίμα και την ενέργεια. Διότι ναι μεν στα ενεργειακά η βιομάζα θα έπρεπε να ανέβει, αλλά η ανησυχία που έχουμε είναι ότι αν ανέβει εκθετικά τότε θα υπάρχει πρόβλημα με τα αιωρούμενα σωματίδια και τους σχετικούς ρηπαντές. Οπομένως πρέπει να βρεθεί μια μέση οδός στην οποία θα λέμε ναι μεν δράσεις για το κλίμα, αλλά πρέπει να είμαστε και βέβαιοι ότι δεν θα πάμε προς την αντίθετη κατεύθυνση και θα δημιουργήσουμε ένα νέο πρόβλημα. Για τον υδράργυρο. Ε, είναι η μόνη ε, προετοιμασία και ε, θα κάνουμε και μια νέα πρόταση σύντομα για το θέμα αυτό. Αναφέρθηκα στην ευελιξία, ίσως θα έπρεπε να πω και δύο λόγια παραπάνω για την οδηγία για τις ε, εθνικές εκπομπές ατμοσφαιρικών ρήπων, διότι σας είπα εν συντομία στην εισαγωγή μου ότι, για παράδειγμα, κάποια κράτη-μέλη ε, έχουν μεγάλες εκπομπές οι οποίες είναι από θαλάσσιες μεταφορές. Αυτές θα μπορούσαν να ξεκινήσουν ε, και να είναι λιγότερο δαπονερές με παραγωγή η οποία θα είναι χερσαία πλέον. Υπάρχει ευελιξία. Ε, για το μεθάνιο, το γεγονό ότι δεν συμπεριλήφθη. Ε, Καταρχά, μπορεί να υπάρχει κοινή εφαρμογή. Αν δύο ή τρία κράτη-μέλη αποφασίσουν ότι είναι φθηνότερο σε ένα κράτος μέλος ε, να το εφαρμόσει ένας ε, αντί για δύο ή τρεις, τότε μπορεί να υπάρξει συμφωνία και να γίνει παραγωγή στη λιγότερο δαπονερή περιοχή. Και όσον αφορά το κόστος, επειδή πολύ συχνά μας ρωτάτε, όχι, δεν είναι δαπανηρό, ε, μας ε, προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία να εφαρμόζουμε αυτές τις επιλογές μηδενικού κόστους οι οποίες υπάρχουν, οδηγούν σε ωφέλη και δεν έχουν κάποια επιπλέον επιβάρυνση. Κάτι τώρα διότι έγινε κάποια αναφορά σε διοικητικό άχθος, ότι κάθε χρόνο γίνονται πλέον μετρήσεις, ότι ε, σε 10, για 10 χρόνια θα πρέπει να αποθηκεύονται τα στοιχεία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνεται αυτή η διαδικασία, διότι αλλιώς δεν μπορούμε να έχουμε κατάλληλες αξιολογήσεις. Αν δεν υπάρχει συνεχής καταμέτρηση των εκπομπών, είναι πολύ δύσκολο κάποια στιγμή να κατανοήσουμε σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο η πρόοδος επετεύχθη και κατά πόσον αυτή συμμορφούνται με τους στόχους μας. Αυτό είναι ακριβώς το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Και φυσικά η ανάλυση ε, ε, δεν θα είναι και τόσο ε, καλή εάν δεν έχουμε λιγότερα στοιχεία. Ναι, υπάρχει κάποια διοικητική επιβάρυνση, αλλά είναι πολύ μικρότερη σε σχέση με τα ωφέλη τα οποία έχουμε από τη συγκεκριμένη πρόταση. Και Εσκεμένα ε, στις μεσαίου μεγέθους μονάδες κάσις, έχουμε συμπεριλάβει ε, και ε, κάτι το οποίο προβλέπεται για τις μεγάλες ε, ε, μονάδες καύσης, διότι θεωρήσαμε ότι δεν ήταν απαραίτητο να έχουμε πλήρη καταμάφραση. Γίνεται μία απλώς ε, εγγραφή και το κόστος μειώθηκε από τα 20 εκατομμύρια στα 9 εκατομμύρια. Ναι, υπάρχει ακόμα κάποιο κόστος, αλλά είναι το ελάχιστο δυνατό και θεωρούμε ότι μπορούμε να εξισορροπήσουμε το κόστος αυτό με τα ωφέλη. Ελπίζω να απάντησα σε ε, περισσότερες από τις ερωτήσεις, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες τις παρατηρήσεις σας και όλα τα σχόλιά σας. Θα ήθελα να ζητήσω από τους κοιότης μας και τους δύο να ολοκληρώσουν και να συνοψίσουν τη συζήτηση. Να παρακαλέσω πρώτα τον κύριο Άνταμ Γκέρεκ που είναι ο συντάκτης γνωμοδότησης για την πρώτη πρόταση οδηγίες που αφορά τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρήπων. Κύριε Γκέρεκ, παρακαλώ. Στις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν βλέπουμε πολλές ενδείξεις ότι η τελευταία πρώτος οδηγίας είναι σημαντικότερη από τις προηγούμενες για το διοξίδιο του άνθρακα. Έτσι φαίνεται, αλλά η, η, η επιρροή στις κλιματικές αλλαγές σίγουρα θα είναι τεράστια, τεράστια, αλλά θα ήθελα να σας υπενθυμίσω και πάλι το θέμα των ε, πολύ επικίνδυνων ε, αιωρούμενων σωματιδίων, των πολύ μικρών, που έχουν νανομετρικά μεγέθη, δηλαδή διάμετρο κάτω από 2,5 ε, εκατομμυριστό του μέτρου. Αυτά δεν περιλαμβάνονται. Είναι βέβαια τεράστια πρόκληση για αυτούς που πρέπει να κάνουν τη μέτρηση, αλλά από την άλλη πλευρά αυτή, αυτά τα αιωρούμενα σωματίδια είναι ένα σημαντικό μια σημαντική αιτία των κλιματικών αλλαγών. Γιατί λοιπόν η οδηγία δεν λαμβάνει υπόψη και αυτά τα πολύ μικρά αιωρούμενα σωματίδια, ίσως θα μπορούσε να τροποποιηθεί από ε, αυτού. Βέβαια, δεν μπορούμε ακόμη να προσδιορίσουμε ε, τις, ε, το σύνολο των εκπομπών αυτών των μικρών αιωρούμενων σωματιδίων, αλλά τουλάχιστον να μιλήσουμε για τις πηγές εκπομπών για να δούμε αν μπορέσουμε τις πηγές να μειώσουμε ή να εξαλείψουμε. Δυστυχώς δεν βλέπω στην πρώτη οδηγίας ε, μέτρα δράσης. Μιλήσατε για τον ντίζελ. Με ποιο τρόπο θα επηρεάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ε, εκπομπή αξιδίων του αζότου που προκαλούν ε, φθορά του, του στρώματος του όζοντος γιατί γνωρίζουμε και έχουμε κάνει τη διάγνωση ότι επηρεάζει το όζον και τα διοξίδια του αζότου τις κλιματικές αλλαγές, αλλά πώς μπορούμε να επηρεάσουμε την, τις εκπομπές δίζελ. Θα περιορίσουμε την κυκλοφορία των, ε, αυτοκινήτων. Πρέπει να έχουμε κάποια συμφωνία ε, με, τους, ε, με την αυτοκινητοβιομηχανία σε τέτοια περίπτωση. Αλλά δεν βλέπω εδώ δυνατότητες επιρροής της κατάστασης. Αυτό λείπει στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ωραία, θα δώσω τώρα το λόγο στο συντάκτη γνωμοδότης της δεύτερης πρότασης ε, που αφορά τα μεσαία μεγέθους μονάδες κάψη, ο κύριος Φέντελε. Ήταν καλή η παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και νομίζω ότι ήταν ε, καλή συζήτηση που έγινε με τους συναδέλφους από τις πολιτικές ομάδες. Έχω την αίσθηση πάντως ε, ότι θα έχουμε μεγάλη διαφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την εφαρμογή αυτής της οδηγίας. Βέβαια είναι αναφυσβήτητο ότι έχουμε κάποια εμπόδια που θα πρέπει να τα υπερκεράσουμε. Γιατί έχουμε πραγματικά πολύ σημαντικό τομέα. Η ενέργεια είναι κέριο ζήτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά θα πρέπει να ακούσουμε και τα επιστημονικά πορίσματα και να λάβουμε υπόψη και το κόστος για την κοινωνία αλλά και την επίδραση στην δημόσια υγεία. Και όταν μιλάμε για τη σχέση κόστους-οφέλους, στον υπολογισμό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα δεινά των ανθρώπων που αρρωσταίνουν, που υποφέρουν, για να μην μιλήσουμε για την επιβάρυνση στα συστήματα υγείας και το σχετικό κόστος. Έχουμε λοιπόν και θέμα δημόσιας υγείας και οικονομικό ζήτημα. Όλα αυτά θα πρέπει να εξετάσουμε από κοινού και θα το συζητήσω με τους συναδέλφους από τις άλλες ομάδες. Σας ευχαριστώ κύριε Φέντερλε. Πλησιάζουμε προς το τέλος ε, της συζήτησης, κυρία Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, που είστε αρμόδια και για τα δύο θέματα. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συζήτηση. Θα τα ξαναπούμε στο μέλλον. Σας ευχαριστώ, συνάδελφοι. Λύεται η συνεδρίαση, εκτός και αν έχετε καμιά πρόταση για τα διάφορα. Έχετε τίποτα στα διάφορα. Όχι. Σας ευχαριστώ. Ραντεβού τη Δευτέρα στην πρώτη ακρόαση. Καλή σας ημέρα.